So, Κυρίες και κύριοι, νομίζω πως είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Κάτι υπάρχει ηχό μέσα στην αίθουσα, δεν ξέρω τι φταίει. Δεν έχει κανείς άλλο στο μικρόφωνο ανοιχτό. Τέλος πάντων, έλεγα πάλι πως ε, συνεδριάζουμε σε αυτή την σπηλαιώδη αίθουσα και υπάρχει ηχό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει... έχει περάσει πολύ καιρό από την τελευταία μα συνεδρίαση λόγω του χρονοδιαγράμματο του Κοινοβουλίου. Σα καλωσορίζω λοιπόν. Ω συνήθω μεταδιδόμαστε στο διαδίκτυο. Καλά δεν λέω. Καλωσορίζω λοιπόν και οποιονδήποτε μας παρακολουθεί στο διαδίκτυο. Να σας υπενθυμίσω επίσης πως ε, προσθέθηκαν ε, εδώ πέρα νέα ενημερωτικά δελτία της Επιτροπής μας. Έχουμε μία συλλεκτική θα την έλεγα έκδοση για το φόρουμ της ενιαίας αγοράς στην Κρακοβία και για την οποία ευχαριστώ τον Φρεντερίκο και την ομάδα που συμπεριλαμβάνει και τη διακήρυξη της Κρακοβίας και μετά έχουμε την έκδοση του Νοεμβρίου που έχει έτσι ένα πιο ωραίο εξώφυλλο με τα θέματα μέσα σε κουτάκια. Βλέπετε εδώ πέρα νέες ιδέες. Οπότε έχετε και αυτά να δείτε. κατόπιν. Έχουμε τα πρακτικά της 26 ης Σεπτεμβρίου που έχουν υποβληθεί. Αν έχετε κάποιο σχόλιο, παρακαλώ, πριν το τέλος συνεδρίασης να μου το πείτε. Ε, το τέλος εννοώ την Τετάρτη βεβαίως, αλλιώς θεωρώ πως έχουν εγκριθεί. Επίσης, ε, θα ήθελα να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη και να σας πω πως υπάρχει άλλη μια αλλαγή στην ημερήσια διάταξη γιατί ε, ειδικά η κυρία Γκέπχαρτ θα αναχωρήσει για τη Δανία αυτή την εβδομάδα οπότε προτείνουμε οι συντονιστές να συνεδριάσουν αύριο στις 11 η ώρα από τις 11 μέχρι τις 12.30 και μετά νομίζω το θέμα της κυρίας Γκέπχαρτ ε, θα είναι πρώτο πρώτο τρίτη πρωί και μετά το θέμα Πέρες θα πάει την Τετάρτη. Αλλάξατε δηλαδή μεταξύ σας. Ωραία. Αλλά ειδικά για τους συντονιστές πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα. Οπότε, εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Ωραία, να σας υπενθυμίσω πως τρίτη απόγευμα έχουμε την ακρόαση Κρόιτσμαν για την ε, προστασία καταναλωτών και εργατικά δικαιώματα και την ε, περί Οπότε ενημερώστε τις ομάδες σας για να έχουμε μεγάλη παρουσία βουλευτών. Αυτές νομίζω είναι όλες οι ανακοινώσεις. Οπότε, τώρα θα περάσουμε στο πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης. που είναι μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας για τον πίνακα αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς και καλωσορίζω τον Σάιμον Μπουσουτή, που θα είναι ο εισηγητής και μετά έχουμε τον κύριο Κορέα Ντεκάμπος, ο κύριος Λόχιγκερ αποσιάζει, ξέρω πως ο κύριος Κρόιτσμαν θα τον απληρώσει, κυρία Ρούλε αποσιάζει, εγώ θα εκπροσωπήσω το ECR, οπότε ελπίζω κάποιοι να βρεθούν να συζητήσουν μαζί σας. Αλλά θα έχετε ενδιαφέροντα πράγματα οπωσδήποτε. Και να δούμε ποιος είναι εδώ πέρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όχι, κανείς. Κάποιος θα έρθει, είμαι σίγουρος. Ωραία. Ευθύς αμέσως λοιπόν. Δεν ξέρω, υπάρχει κανείς από την Κομισιόν. Όχι. Σάιμον, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι ευχαρίστηση για μένα η ευθύνη να ασχοληθώ με την έκθεση αυτή για τον πίνακα βαθμολογίας της εσωτερικής αγοράς. Ξέρετε πως στην ενδιάμεση περίοδο μέχρι να μπει στην ημερήσια διάταξη το θέμα αυτό έχει δημοσιευτεί η 23η έκθεση και άρα η δική μου η έκθεση θα δει και την 22η και την 23η έκθεση. Και βεβαίως πρόκειται για μια ιδιαίτερη χρονική στιγμή όπου όλοι εδώ στο Κοινοβούλιο και εκτός συζητάμε το τι συμβαίνει στην Ευρωζώνη και η έκθεση αυτή μας δίνει την ευκαιρία να εξετάσουμε ένα από τα πιο σημαντικά τι πιο σημαντικές πτυχέ αν όχι την πιο σημαντική πτυχή τη Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση που είναι η ενιαία αγορά και βεβαίω είναι η δυνατότητα που έχουμε, ειδικά στην κατάσταση που είμαστε, για να ανακτήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο κάναμε από κοινού, έχει λειτουργήσει και ελπίζω θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε. Και ο πίνακα αυτός βαθμολογίας βεβαίως πηγαίνει ειδικά προς αυτή την κατεύθυνση με το να δημοσιεύει το τι κάνει το κάθε κράτος μέλος, το πόσο καλά τα πηγαίνει όσον αφορά την εφαρμογή της εσωτερικής αγοράς. Η έκθεσή μου, κύριε Πρόεδρε, κατ' ουσίαν αφορά τρία πράγματα. Πρώτα απ' όλα βεβαίως, τους πίνακες αυτούς που ανέφερα, μετά το Solvit, γιατί ε, και αυτή η έκθεση θα ε, ενταχθεί στην δική μου κατόπιν θα δούμε τρόπους να επιτύχουμε τον κοινό στόχο βελτίωσης ε, της εφαρμογής και της επιβολής των κανόνων της κοινή αγοράς και τρίτον όσον αφορά την απόδοση των προβλημάτων δικτύων λύσεως προβλημάτων όπω το Solvit. Δεν ξέρω αν είναι σύμπτωση, αλλά βεβαίω εγώ κατάγομαι από μια χώρα η οποία έχει βαθμολογηθεί ως η χώρα με την καλύτερη εφαρμογή των κανόνων της εσωτερικής αγοράς. Η χώρα μου, η Μάλτα, είναι αυτή η οποία έχει κάνει την καλύτερη, την πληρέστερη εφαρμογή. Δεν ξέρω εάν ε, γι' αυτό μου έδωσε αυτή την έκθεση ο συντονιστής μου, αλλά ευχαρίστως βεβαίως ε, λαμβάνω αυτή τη δουλειά για να δείξω πως είναι πράγματι δυνατόν να προχωρήσουμε, να εφαρμόσουμε και να συμμορφωθούμε με τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει τα κράτη-μέλη στο επίπεδο της Ένωσης. Κύριε Πρόεδρε, δεν θέλω τώρα να μείνω στις λεπτομέρειες της έκθεσης της ίδιας. Περίμενα να είναι εδώ η Κομισιόν για να τις παρουσιάσει, φαίνεται πως δεν είναι εδώ, αλλά θα αναφέρω την προσέγγιση που θα ακολουθήσω. Και βεβαίως ευχαρίστως να ακούσω και τους συναδέλφους. Πρώτα απ' όλα λοιπόν θα ήθελα η έκθεση να τονίσει την σημασία της μεταφοράς ε, της κοινοτικής νομοθεσίας ε, με τρόπο έγκαιρο και αποτελεσματικό. Θα ήθελα να τονίσω, κύριε Πρόεδρε, πως ε, από την θέση ενισχύ τη συνθήκης της Λισαβόνας 1 Σεπτεμβρίου 2009 το δικαστήριο της Ένωσης για πρώτη φορά είχε δυνατότητα να επιβάλλει πρόστιμα αμέσως εάν τα κράτη-μέλη δεν είχαν εκπληρώσει τα καθηκόντά τους όσον αφορά την μεταφορά στο εθνικό δίκαιο ε, οδηγιών. Και θα ήθελα να μας πει η Κομισιόν ε, ε, εάν ε, έχει γίνει τίποτα σε σχέση με το άρθρο 260 παράγραφος 3. Κατόπιν έχουμε την σημασία του Ευρωπαϊκού Δικαίου και την σημασία της σωστής εφαρμογής του, καθώς σε πάρα πολλές περιπτώσεις αντιμετωπίζουμε καταστάσεις οποίες τα κράτη-μέλη δεν μεταφέρουν ε, επαρκώς την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και αυτό προφανώς δημιουργεί δυσκολίες στη φάση της εφαρμογής. Και βεβαίως θα τονίσω την σημασία της σωστής εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και μια ισχυρότερη ιστορική αγορά. Κύριε Πρόεδρε, συνήθως στους νόμους, στη ρύθμιση, τη νομοθεσία τα θεωρούμε γραφειοκρατία. Αυτό το οποίο θα προσπαθήσω εγώ να πω είναι πως η ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας έχει ωφέλη για τις επιχειρήσεις, για τους πολίτες και άρα δημιουργεί μια ισχυρότερη εσωτερική αγορά. Αυτά. Θα σταματήσω λοιπόν εδώ πέρα στη, τη σύντομη εισαγωγή μου. Αναμένω βέβαια στους απόψεις των συναδέλφων και βεβαίως ε, την συνεργασία με τους συναδέλφους και τους σκιώδεις συζήτητες Αναμένουμε λοιπόν μια πρώτη συνάντηση για να ανταλλάξουμε απόψεις και να μπορέσουμε να έχουμε μια έκθεση η οποία θα βασίζεται ε, σε μια συνένεση για να μπορέσει να ευθετηθεί τις ερχόμενες εβδομάδες. Ευχαριστώ, Σάιμον δίκαιο έχετε που υψημένετε αυτά τα οποία έχει επιτύχει η Μάλτα και νομίζω πως ήταν ένας λόγος για τον οποίο αναλάβατε αυτή την έκθεση γιατί νομίζω πως ε, έχετε άρα έτσι, ένα ηθικό ανάστημα και μπορείτε να, να διδάξετε κάποια πράγματα και αναμένουμε τις ε, απόψεις Θα επανέλθω κι εγώ αργότερα. Τώρα οι σκιώδεις συζήτητες. Καλωσορίζω την κυρία Ρούλε, η οποία βλέπω πως είναι σκιώδης. Δεν ξέρω αν το ξέρατε. Ο καθηγητής ο Κορέαντε Κρόιτσμαν, Ρούλε και μετά θα μιλήσω εγώ για την ομάδα μου και αν θέλει κάποιος άλλος να μιλήσει. Ε, Ευχαριστώ. Οπότε κύριος Κορέντε Κάμπος. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τον συνάδελφο Μπουσουτήλ για διάφορους λόγους. Ένας εξ αυτών είναι ότι Ακριβώς είναι ένα από τα λίγα άτομα που δεν έχει σύγκρουση φερόντων σε αυτή την υπόθεση και θα ήθελα να συγχαρώ και τη χώρα του σε αυτό το τομέα. Συμφωνώ δε και με τα σχόλια που διατύπωσε και είναι σχόλια επί των οποίων ε, περισσότεροι από εμά συμφωνούμε. Ο αριθμός των παραβάσεων είναι πολύ μεγάλος. Ο αριθμός δηλαδή το Ισμή μεταγραφής οδηγιών είναι τεράστιος. 90 οδηγίες δεν έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα λόγω το Ισμή μεταγραφής τους από κάποια κράτη-μέλη. Για μας αυτό σημαίνει αρκετά χρόνια δουλειάς. Γι' αυτό και προκύπτει αυτή η ιδέα ότι πρόκειται για απώλεια της ε, πνευματικής μας παραγωγής που θα έπρεπε να αποφεύγεται. Υπάρχει όμως και μια θετική πτυχή. Ε, ενώ έχουμε 25% λιγότερες παραβάσεις φέτος και έχουμε και άλλες δεσμεύσεις μέχρι Έχουμε και άλλε μάλλον δεσμεύσει για άλλα κεφάλαια και άλλου τομεί. Η ανησυχία μου βασικά και η συμβολή μου για αυτή την έκθεση είχε να κάνει με το πώς θα μπορέσουμε να μειώσουμε τις προθεσμίες και τον αριθμό παραβάσεων και καθυστερήσεων στη μεταγραφή Θεωρώ πως ο βασικός στόχος αυτών των πλαισίων είναι να επιστήσουμε την προσοχή κάθε χώρας με κομψό μεν τρόπο αλλά και επιτακτικό ταυτόχρονα και πιστεύω πως εδώ εμείς οι ευρωβουλευτές έχουμε ένα ρόλο να παίξουμε. Εγώ ήδη είχα εντατικές επαφές με τους αρμόδιους της χώρας μου προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να επιστήσω την προσοχή τους όταν θεωρώ πως ε, τα αποτελέσματα δεν είναι πολύ καλά. Από την άλλη πλευρά είναι ένας τομέας όπου μπορούμε να συνεργαστούμε με τους ε, εθνικούς βουλευτές. Δεν ξέρω τι πιστεύει ο Πρόεδρος, αλλά έχουμε ήδη επαφές με τα εθνικά κοινοβούλια και γι' αυτό ίσως θα άξει τον κόπο να έχουμε την υποστήριξή τους σε αυτή την υπόθεση. Ε, εν πάση περιπτώσει να τους ενημερώσουμε και να τεθεί αυτό το θέμα στη συζήτηση κάθε ε, φορά που έχουμε επαφές. Κατά τα άλλα δεν έχω διαφορές με τον ε, συνάδελφο Τίλε. Εσπέρα πως θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε και στο μέλλον για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κρόιτσμαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εξ ονόματο συναδέλφου Λούντριγκάρτα θα ήθελα να σα κάνω κάποιε συστάσει για αυτό το θέμα. Είναι κέρια η έκθεση γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται περισσότερο από ποτέ ομαλά λειτουργούσα εσωτερική αγορά που θα οδηγήσει σε ανάκαμψη της οικονομίας και περισσότερες θέσεις απασχόλησης, καθώς και θα αυξήσει την αγοραστική δύναμη των Ευρωπαίων πολιτών. Πολλά ήδη έχουν γίνει, ωστόσο μόνο τα 11 κράτη-μέλη έχουν επιτύχει το κατόφλι του 1%. Μείωση από το 20% πέρυσι ε, μάλλον τα περασμένα χρόνια. Σημαίνει πως, πρέπει να, ε, πως μειώνονται έτσι οι επιλογές για τη βελτίωση της οικονομίας. Μια σωστά λειτουργούσα οικονομία είναι το κλειδί για τη σωστά λειτουργούσα ευρωπαϊκή οικονομία. Τώρα είναι λοιπόν η κατάλληλη στιγμή τα κρατημέλη να επιταχύνουν τις προσπαθειές τους για να μεταγράψουν ορθά και έγκαιρα τις ε, οδηγίες σε νομοθεσία δική τους. 16 κράτη-μέλη είναι πάνω από το 1%, το κατόφλι του 1%. Δεύτερον, τα κράτη-μέλη θα έπρεπε να εφαρμόζουν τις οδηγίες ε, ε, άμεσα. Ε, επιπλέον, ε, πολλές οδηγίες δεν, είναι, δεν εφαρμόζονται σωστά και δεν είναι ντροπή να επαναλαμβάνουμε ένα καλό επιχείρημα ή να επαναλαμβάνουμε μια καλή ιδέα που έχει δοκιμαστεί παλιότερα. Δηλαδή, η να επαναλαμβανουμε μια καλη ιδεα που εχει δοκιμαστει παλιοτερα δηλαδη αυξηση της ενημέρωσης για την ε, ελλειπή εφαρμογή και μεταγραφή των οδηγιών. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω της ενημέρωσης του κοινού και μέσω της πίεσης ε, από τους υπολείπους. Χρειάζεται λοιπόν να ξεκινήσει μια ε, πιο ευανάγνωστη μορφή του πίνακα επιδόσεων των κρατών μελών για την εσωτερική αγορά, έτσι ώστε να ενημερωθεί ευρύτερα το κοινό και έπειτα όταν θα ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια ε, να γίνει γνωστό, να δημοσιοποιηθεί περισσότερο για να, και να δημοσιοποιηθούν και οι επιπτώσεις των παραβάσεων. Αυτά ήθελα να τονίσω. Σας ευχαριστώ. Uh, thank you Κυρία Ρούλε, ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομη. Συμφωνώ με του προλαλήσαντες. Δεν θα τα επαναλάβω. Να αναφέρω κάτι το οποίο θα μπορούσε να παίξει ένα ρόλο στην έκθεση. Η Επιτροπή μας κάνει συνεχώς εκθέσει ίδιες πρωτοβουλίε για την εφαρμογή και τη μεταφορά των οδηγιών. Θα μπορούσε λοιπόν ο εισηγητή που ε, επεξεργάζεται τον πίνακα βαθμολογίας να ε, μπορέσει να μας πει σε τι θα μπορούσαμε να δώσουμε ιδιαίτερο βάρος. Αλλιώς συμφωνώ πλήρως με τις προτάσεις του κυρίου Μπουστήλ και αναμένω τη συνεργασία μας. Ναι. Εκ μέρου της δικιά μου ομάδα τώρα. Παρακολουθούμε αυτό το τομέα από κοντά. Η έκθεση αυτή πιστεύω ότι είναι μια σημαντική έκθεση. Είναι βέβαια μια προσωρινή έκθεση, μεταβατική. Δεδομένου ότι υπογραμμίζουμε πάρα πολύ από την ενία πράξη το θέμα της ε, προσαρμογής της εθνικής νομοθεσίας στην ε, ευρωπαϊκή. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και την οδηγία για τις υπηρεσίες. Φαντάζομαι θα προχωρήσουμε και εκεί. Η έκθεση αυτή λοιπόν πιστεύω ότι είναι προς το παρόν αρκετά πλήρης, αξιόλογη, δίνει νέο υλικό, κάτι το οποίο είναι πολύ θετικό. Συνεπώς, φέτος η έκθεση αυτή αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία γιατί πρέπει να προσπαθούμε να προσφέρουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή νέες ιδέες. Η ενιαία αγορά έχει πολλούς ειδικού ε, στόχους, το υπογραμμίζουμε αυτό. Και τώρα ένα από τα πράγματα τα οποία ίσως θα έπρεπε να δούμε είναι μήπως τελικά έχουμε υπερβολικά πολλές εκθέσεις και θα έπρεπε να τις συγκεντρώνουμε κάπως και να δούμε πώς συνδέονται μεταξύ τους. Για το Solvit, για παράδειγμα, υπάρχει συσχετισμός ανάμεσα στα προβλήματα τα κυριότερα στο Solvit και αυτά τα οποία αντιμετωπίζουμε εμείς όταν εξετάζουμε τη λειτουργία της ενίας αγοράς. Έχουμε όμως κάποιες αρχές, τις οποίες θέλουμε να σεβαστούμε απέναντι στους πολίτες. Έτσι λοιπόν, Η κάθε έκθεση που θα ετοιμάσουμε πρέπει να επικεντρώνεται περισσότερο στον πολίτη. Ενώ μέχρι τώρα ίσως το κάνουμε περισσότερο προς την έρευνα και λιγότερο κατευθύνουμε τις εκθέσεις μας προς τους πολίτες. Θα έπρεπε να έχουμε πιο στρατηγική σημασία σε εκθέσεις τώρα από ό,τι κατά το παρελθόν. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από τον εισηγητή να πάει προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτά έχω να πω εγώ. Τώρα, ο Hans Peter Mayer και δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι που θέλουν να πάρουν το λόγο. Ας ακούσουμε τον Hans Peter και μετά έχουμε χρόνο αν κάποιος θέλει κάτι να προσθέσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συζητάμε εδώ πέρα βέβαια. Θα συζητήσουμε σε λίγο για το πρόγραμμα εργασίας της Κομισιόν. Άρα γίνεται ακόμη πιο σημαντική έκθεση του κυρίου Μπουσουτήλ. να υπενθυμίσω πως μιλάμε για την εφαρμογή. Εμείς μπορούμε να αποφασίζουμε ότι θέλουμε, αλλά δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα εάν δεν εφαρμοστεί και δεν εφαρμοστεί σωστά. Δύο σύντομα παραδείγματα. Πρώτον, εδώ και δύο χρόνια έχουμε ενισχύει μια διαδικασία περί μικρών διαφορών, δηλαδή μέχρι 2.000 ευρώ μπορεί κανείς γρήγορα να ζητήσει αποζημίωση ή οτιδήποτε στην πράξη δεν γίνεται τίποτα. Ενδιαφέρθηκα να δω μία περίπτωση από τη δική μου την περιφέρεια και τι έγινε. Εκεί πέρα πράγματι εντός εξαμήνου όπως ε, ε, προβλεπόταν ε, αποζημιώθηκε ο επιβάτης γιατί επρόκειτο για μια αεροπορική εταιρεία, με ένα ταξίδι προς την Ολλανδία και η εταιρεία βεβαίω ε, είχε έδρα επίσης στην Ολλανδία και είχε υποκατάστημα στη Γερμανία οπότε προσέφυγε στο τοπικό δικαστήριο ο ενδιαφερόμενος και είχαμε γρήγορα ε, αποτέλεσμα στην Ολλανδία μέσα σε έξι μήνες. Πριν Είχε προσπαθήσει ο άνθρωπος, του λέγανε πρέπει να πας στην Ολλανδία, ο Ολλανδός δικηγόρος θέλει 2.000 ευρώ προκαταβολή. Οπότε λέει το ξέχασέ το. Οπότε η όλη διαδικασία ε, είχε κόστος 590 ε, ευρώ τους ή άλλους, τα οποία ε, πληρώθηκαν. Οπότε έχει εφαρμοστεί, αλλά έχει μεταφερθεί, με συγχωρείτε, αλλά δεν εφαρμόζεται γιατί δεν το ξέρουν ακόμα καν τα δικαστήρια. Αυτό είναι θέμα οργάνωση των κρατών μελών, όχι του λαού. Πρέπει να, να ενημερωθούν. Αν δεν το ξέρουν ούτε οι δικαστέ, δεν έχει κανένα νόημα. Και δεύτερον, ποιο είναι το πρόβλημα τώρα. Έχουν πρόβλημα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ειδικά όσον αφορά τον τομέα της γεωργίας. Έχουμε τώρα μία νομοθεσία ε, όσον αφορά τα πουλερικά όπου θα πρέπει από 1η 1η 2012 να έχουν κάποια ειδικού, ειδικούς διαμορφωμένους ε, κλωβούς για τις ε, κότες οι οποίες κάνουν αυγά. Μιλάμε για ένα 20% των επιχειρήσεων σε Αυστρία και Γερμανία που έχουν συμμορφωθεί με μεγάλο κόστο. Προσπάθησε η Κομισιόν να το εφαρμόσει και στι υπόλοιπε. Δεν συνέβη τίποτα. Τι θα γίνει λοιπόν τώρα. Σε δύο μήνε από πρώτη πρώτου, ε, τι γίνεται. Είμαστε σε μία αγορά. Κάποιοι άνθρωποι λοιπόν θα έχουν υψηλότερο κόστος και αυτοί οι οποίοι παρανομούν πλέον από πρώτης πρώτου θα είναι φτηνότεροι. Οπότε ζητάμε εδώ πέρα και έχουμε μία διακήρυξη για να απαγορευτούν τα αυγά τα οποία δεν προέρχονται από τις ε, υπόλοιπες εκμεταλλεύσεις. Βεβαίως δεν θα μπορέσουμε να τα απαγορεύσουμε γιατί τα αυγά είναι τα ίδια με αυτά τα οποία παράγονται σήμερα. Δεν είναι ούτε καλύτερα ούτε χειρότερα. Απλά έχει αλλάξει η νομοθεσία. Μάλλον τα κλουβιά δηλαδή Επίσης μην ξεχνάμε πως εξακολουθούμε να εισάγουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυγά, οπότε δεν έχει νόημα να το απαγορεύσουμε αυτό. Αλλιώς θα σταματήσουμε να παράγουμε ζυμαρικά. Οπότε πρέπει να δούμε όταν εφαρμόζουμε κάτι να εφαρμόζεται παντού. Δεν είναι δυνατόν να μας ε, ξεφεύγουν τέτοια πράγματα και μετά να έχουμε την επόμενη οδηγία ακόμη αυστηρότερη για την ευζοία των ζώων, των ανθρώπων και ξέρω εγώ πιανού και να μην γίνεται τίποτα. Μέχρι και αυτοί οι οποίοι τώρα δεν κάνουν τίποτα να κάνουν, δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουμε παραπέρα. Οπότε αυτή η έκθεση είναι πάρα πολύ σημαντική και είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα η πλήρης ε, μεταφορά και εφαρμογή του κοινωτικού δικαίου και στις 27 χώρες. Uh, είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λέτε. Το συζητήσαμε όταν ήμασταν και στους πίνακες συσχετισμών. Τώρα, ποιος άλλος θέλει το λόγο. κύριος Σβάπ είναι επόμενος στο καταλογό μου. Ε, κύριος ευχαριστώ μετά από αυτά ε, τα οποία είπε ο κύριος ε, Peter ε, θα πρέπει και εγώ βεβαίως να πω πως ε, και για τη δική μου περιφέρεια θα είναι δράμα αν δεν έχουμε αυγά για να φτιάξουμε σπέτς λέει το ζυμαρικό μας εκεί. Τώρα, ο Σάιμον Μπουζουτήλ νομίζω συνεισφέρει σημαντικά στη συζήτηση που είχε ξεκινήσει με τον ε, Μάριο Μόντι ε, ο οποίος είχε παρουσιάσει το σχετικό του έγγραφο στην Επιτροπή μας, οπότε θα πρέπει να έχουμε μόνο μια οικονομική διακυβέρνηση, αλλά και μια διοίκηση της εσωτερικής αγοράς. Και οπωσδήποτε η έκθεση αυτή συνεισφέρει σε αυτό, αλλά είναι μια έκθεση η οποία ήταν στατική και εδώ πέρα έχει δίκιο ο Χανς Πέτερ Σμαέρ και κοίταζε το εάν ε, υπήρχε εφαρμογή, το εάν υπήρχε όντως ορθή και πλήρης ε, χρήση είναι κάτι το τελείως διαφορετικό. Και τέλος, το ανέφερε και αυτό και ο πρόεδρος, θα πρέπει η έκθεση αυτή να συνδεθεί και με άλλα στοιχεία παρακολούθησης, εφαρμογής των οδηγιών. Ε, είπατε τους ε, πίνακες συσχετισμού, πολύ σωστά κύριε Πρόεδρε, αλλά νομίζω πως χρειάζεται να γίνει και μια συζήτηση για το πώς θα καταφέρουμε να εξετάσουμε την αποτελεσματικότητα βεβαίως των θεσμικών οργάνων για να δούμε μήπως ε, χρειάζεται περισσότερους κανονισμούς η κοινότητα για να έχουμε μια πιο γρήγορη διαδικασία. Οι διαδικασίες επί παραβάση μέχρι στιγμής αφορούν ε, την μη εφαρμογή αλλά σπάνια την μη επαρκή ε, εφαρμογή. Οπότε η Κομισιόν με το πακέτο αυτό το οποίο πρότεινε πριν από δύο εβδομάδες νομίζω θα συνεισφέρει αρκετά και εμείς ως Κοινοβούλιο θα πρέπει να τη στηρίξουμε. Ευχαριστώ. Άλλοι δύο είναι στο καταλαγό μου, Σαλτεμόσα και Βάιλερ. Και μετά θα δώσω το λόγο στον κύριο Μπουσίτελ για να συνοψίσει. 3 και 45 κανονικά πρέπει να αρχίσουμε την ψηφοφορία ε, που θα είναι σύντομη για την επόμενη γνωμοδότηση που πρέπει σήμερα να την κάνουμε για να πάει στην επί της ουσίας αρμόδια επιτροπή. κυρία Βαλτεμόση. Ευχαριστώ πρόεδρε. Τώρα που έχουμε χρόνο θέλω και εγώ να πάρω το λόγο για να στηρίξω τους συναδέρφους. Είναι αλήθεια, είναι προφανές ότι υπάρχει ένας καλύτερος τρόπος για να εφαρμόζουμε την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Όσον αφορά τα αυγά, αυτό είναι πρόβλημα και στη Δανία. Να ξέρετε ότι οι καταναλωτές δεν καταλαβαίνουν γιατί πρέπει να είναι τόσο δύσκολο. Έχω λοιπόν μία πρόταση για την Επιτροπή μας και αυτή είναι ότι πέρα από τη στρατηγική που συζητάμε, να καθίσουμε να σκεφτούμε, να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων με το Συμβούλιο για αυτά. Για την αρμοδιότητα των χωρών μελών η εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής. Γιατί λοιπόν να μην προσκαλέσουμε εδώ το Συμβούλιο να έρθει να έχουμε ανταλλαγή απόψεων μαζί τους και έτσι να δούμε μαζί τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να λειτουργεί η ρύθμιση όσο γίνεται καλύτερα. Υπάρχουν διάφορα θέματα, τα τελωνία αλλά και άλλα. Πολλά θέματα που θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε την κατάσταση αν θέλουμε να πείσουμε τον καταναλωτή ότι η ενιαία αγορά είναι κάτι το οποίο όντω λειτουργεί καλά. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Κυρία Βάιλερ. Δυστυχώς φεύγει ο κύριος Μάιερ. Όχι, όχι, δεν είναι μόνο το σπέτσλε το θέμα μας. Ε, κύριε Σφάμπ, πείτε μου εσείς. Καταλαβαίνω βεβαίως αυτό το οποίο αισθάνεσαι αισθάνεστε για την κατάσταση στη Γερμανία σε σχέση με τα ορνηθοτροφία. Αλλά δεν ισχύει ακριβώς... Κοιτάξτε, δεν ισχύει ακριβώς αυτό το οποίο λέτε. Δηλαδή, αναφέρετε ένα παράδειγμα στο οποίο τυχαία η Γερμανία εφάρμοσε κάτι γρήγορα και ορθά. Αλλά ε, για να είμαστε ειλικρινεί, η Γερμανία συχνά δεν τα καταφέρνει πάρα πολλά. Και υπάρχουν κράτη-μέλη, όχι η Δανία, ε, εάν δει κανεί τον πίνακα βαθμολογία που δεν ε, εφαρμόζουν σωστά ή επαρκώς ε, ή εγκαίρως την νομοθεσία. Όλοι νομίζω λοιπόν εδώ πέρα φταίνε, κανείς δεν είναι αναμάρτητος και όπως είπε και η κυρία Σαλτεμόζε έτσι και εγώ θα ήθελα να έχουμε μια στρατηγική συζήτηση με το Συμβούλιο. Οπότε, γιατί τι γίνεται. Ε, το Συμβούλιο είναι εκεί πέρα όταν είναι να λάβει τι αποφάσει. Μετά στην εφαρμογή δεν υπάρχει Συμβούλιο. Και θα ήθελα μια πιο ανοιχτή συζήτηση με τους συναδέλφους στα Εθνικά Κοινοβούλια. Γιατί τουλάχιστον η αντιπολίτευση εκεί πέρα θα μπορούσε να ρωτήσει γιατί δεν εφαρμόζει την νομοθεσία η κυβέρνηση, αν δεν το κάνει η κοινοβουλευτική ομάδα της κυβέρνησης, τότε τουλάχιστον η αντιπολίτευση. Τέλος, έχει δίκιο ο κύριος Μάιερ. Δεν έχει νόημα εδώ πέρα να κάνουμε εμείς ωραίους νόμους και μετά στις χώρες μας να μην λαμβάνονται υπόψη ή να μην εφαρμόζονται πλήρως. Οπότε Έχουμε πάρα πολλά σημεία με τα οποία πρέπει να εργαστούμε Συμβούλιο, Κομισιόν, η Κομισιόν, ο θεματοφύλακας των συνθήκων, θα πρέπει να έχει το θάρρος να πάει τις χώρες στο ΔΕΚ. Αλλά έχουν εντυπώσει πως αυτό συμβαίνει όλο και λιγότερο. Και, και βεβαίως, όπως είπα, και συνεργασία με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Πρόεδρος, Διαπιστώνω και ζητώ συγγνώμη από την Επιτροπή. Υπήρξε ένα πρόβλημα όσον αφορά την ανακοίνωση της ώρας έναρξης της συζήτησης. Ήταν τρεις κανονικά. Δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε. Εν πάση περιπτώσει, τώρα ήρθατε. Χάσατε βέβαια όλη τη συζήτηση για αυτό το θέμα. Αλλά δεν ξέρω αν θέλετε να μας μιλήσετε. Έχουμε την κυρία Φαρχόβεν από την Τίτσι Μάρτε για το βαθμολόγιο. Ποιος από σας θα μιλήσει, παρουσιάστε μας ποιοι είσαστε. Έτσι καλώς είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων που έχουμε για αυτό το θέμα. Ο εισηγητής μας, δίχως άλλο, θα σας μεταφέρει με άλλο τρόπο τα σημεία στο οποίο αναφέρθηκε εδώ. Λοιπόν, ποιος θα ξεκινήσει. Ευχαριστώ. Λέει εκπρόσωπο τη Επιτροπή και ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Όντω, θα σα συστήσω εδώ του συναδέλφου, η κυρία Φερόνικα Καστοκασκάη, η οποία είναι υπεύθυνη για το βαθμολόγιο τη εσωτερική αγορά. Εγώ είμαι η Μανούσκα Γιάνσεν, που είμαι επικεφαλή για το Solvit στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι συνάδελφοι εδώ που βρίσκονται δεξιά μου είναι μέλη τη ομάδα Solvit επίση. Αυτή είναι η ομάδα με την οποία ήρθαμε για αυτό το θέμα. Δεν ήμασταν εδώ βέβαια για να σας ακούσουμε τι είπατε εισαγωγικά Οπότε είναι για μας λίγο δύσκολο έτσι να πάρουμε το λόγο τώρα. Ίσως καλύτερα να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τη συζήτηση και μετά ίσως να παρέμβουμε. Πρόεδρος, εντάξει, την επόμενη φορά όμως που ο κύριος Πουσάτελ θα παρουσιάσει την έκθεσή του, τότε θα πρέπει να έρθετε και να μας ενημερώσετε για τις εξελίξεις. Λοιπόν, θα δώσω το λόγο στον κύριο Μπουσότελ, αλλά προηγουμένω ο κύριο ε, Μα ήθελε πάλι. Γιατί πράγμα για τα αυγά, γιατί σχετικά με την εσωτερική αγορά. Ναι, είναι μια σύντομη παρατήρηση. Όλοι παραπονιόμαστε για το ίδιο πράγμα. Ότι δεν εφαρμόζεται η νομοθεσία και η Κομισιόν και το Συμβούλιο δεν ε, κάνουν τίποτα. Εντάξει, η Κομισιόν μπορεί βεβαίω να πάει τι χώρε στο δικαστήριο, αλλά αφού περάσουν πρώτα απ' όλα οι προθεσμίε. Τώρα για το πράγμα αυτό εδώ πέρα με τις ε, κότες χάρη που θέλαμε πράγματι στα πτυνοτροφία να προστατεύονται τα ζώα. Γνωρίζουμε σε δύο μήνες τελειώνει η μεταβατική περίοδος και γνωρίζουμε πως μόνο 20% ε, έχει υπάρξει εφαρμογή 80% όχι δεν ωφελεί τίποτα μετά την παρέλευση της προθεσμίας να πάμε στα δικαστήρια κτλ. Ε, όταν ξέρουμε ήδη με τις προθεσμίες πως δεν γίνεται τίποτα ε, να μπορούμε να παρεμβαίνουμε. Αυτό πρέπει να σκεφτούμε. Okay. Um... Καλώς. Ωραία. Κύριε Μπουσάντη. Δεν ξέρω όλες τις απειλές βάλτε μαζί. Έχουμε τέσσερα λεπτά μόνο. Ακούγοντα σας θα βοηθηθούν και οι συνάδελφοι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε σας δίνω το λόγο και στο τέλος μιλήστε μας και για το χρονοδιάγραμμα παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ όλους τους συναδέλφους για την βοήθειά τους στη συζήτηση. Την προηγούμενη εβδομάδα ο Επίτροπος Νταλή μου έλεγε ότι είχε πονοκέφαλο με τα αυγά. Τώρα καταλαβαίνω γιατί. Πρόεδρε, Νομίζω ότι το βαθμολόγιο της εσωτερικής αγοράς είναι ένα εξαίρετο εργαλείο, ένα εξαιρετικό μέσο, ένας διπλωματικός τρόπος για να δακτυλοδειχτούμε τα κράτη-μέλη τα οποία δεν στέκονται ε, στην θέση που θα έπρεπε, δεν ε, ενσωματώνουν δηλαδή στην ομοθεσία τους όπως θα έπρεπε το ευρωπαϊκό Δίκιο. Και ακριβώ αυτό πρέπει να γίνεται, να τους δαχτυλοδειχτούμε αν θέλουμε να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα, αν θέλουμε τα κράτη-μέλη πραγματικά να μεταφέρουν στην εθνική τους νομοθεσία ε, τις ε, οδηγίες μας. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο για μια κυβέρνηση κράτους μέλους από το να ε, ακούγονται άσχημα πράγματα γι' αυτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Τσεχία, για παράδειγμα, σήμερα βρίσκεται κάτω-κάτω στο βαθμολόγιο. Παρόλα αυτά, φαίνεται ότι έχει κάνει μία από τις μεγαλύτερες βελτιώσεις ε, τα τελευταία χρόνια σε σχέση με το πίτα στην αρχή. Γιατί, δηλαδή βρίσκεται μεν, έχει το χειρότερο βαθμό στο βαθμολόγιο, από την άλλη μεριά όμως έχει κάνει τεράστια προσπάθεια τελευταία. Να λοιπόν, έτσι αποδεικνύεται η μεγάλη αξία του συστήματος αυτού που έχουμε με το βαθμολόγιο αυτό. Και συνεπώς δεν πρόκειται μόνο για την μεταφορά στην εθνική νομοθεσία, πρόκειται και ίσως και είναι αυτό ακόμα πιο σημαντικό, πρόκειται και για την εφαρμογή της νομοθεσίας, πώς αυτή εφαρμόζεται. Εγώ έρχομαι από μια μεσογειακή χώρα και συχνά οι μεσογειακές χώρες έχουν τη φήμη ότι δεν εφαρμόζουν επαρκώς. Και υπάρχει και κάτι που μπορώ να σας διηγηθώ. ένα ένας επίτροπος για την εσωτερική αγορά μιλούσε με έναν υπουργό μιας μεσογειακής μας χώρας και του έλεγε γιατί δεν εφαρμόζει τους κοινοτικού κανόνες. Και τι είπε, μα τους έχουμε βάλει στον νόμο. Πρέπει και να τους εφαρμόσουμε. Δεν φτάνει που τους έχουμε δηλαδή συμπεριλάβει στην νομοθεσία μας. Βλέπετε, Λοιπόν, η δικιά μου η χώρα που έχει τον καλύτερο βαθμό ίσως μπορεί έτσι να μεταφέρει το μήνυμα ότι ακόμα και οι μεσογειακές χώρες θέλουν και μπορούν να φέρουν σε πέρα τις υποχρεώσεις τους και να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Συνεπώς, η εφαρμογή φυσικά και είναι κάτι πολύ σημαντικό και αυτό θα το συμπεριλάβω στην έκθεσή μου. Έρχομαι τώρα στο χρονοδιάγραμμα, Πρόεδρε. θα συζητήσουμε το σχέδιο έκθεσης στην Επιτροπή μας εδώ τον Ιανουάριο, στις 24 Ιανουαρίου. Έπειτα θα υπάρξει προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου, μέχρι την 21η Ιανουαρίου. Και στη συνέχεια το Φεβρουάριο θα συζητήσουμε τις τροπολογίες και μετά θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας. Είναι από τώρα μέχρι τη συζήτηση του σχεδίου έκθεσης, πάνω από ένα μήνα έχουμε στη διάθεσή μας, Νομίζω ότι μου φτάνει ώστε να συναντηθώ με τους σκιώδεις, όχι μόνο μία φορά, περισσότερες, αλλά να συναντηθώ και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την υπηρεσία και του Solvit και του βαθμολογίου της Επιτροπής, για να είμαστε σίγουροι ότι όσο γίνεται περισσότερο θα είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μια που ο στόχος είναι κοινό μεταξύ μας. Ευχαριστώ και πάλι όλους τους συναδέρφους που συμμετείχαν στην συζήτηση και προσδοκώ σε εξαίρετη συνεργασία μαζί τους. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Μπουσάτιλ. Σίγουρα και οι σκιώδεις συζητητές θα θέλουν πολύ να συζητήσουν μαζί σας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ελπίζουμε οι ιδέες σας να προχωρήσουν. Περνάμε λοιπόν τώρα στο επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη που είναι ψηφοφορία σήμερα για τη γνωμοδότηση όσον αφορά την ε, ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού. Τώρα είμαστε περισσότεροι εδώ, οπότε θέλω να επαναλάβω ότι κάναμε κάποιες αλλαγές της τελευταίας στιγμής στην ημερήσια διάταξη για αύριο. Έτσι, οι συντονιστές θα συνεδριάσουν αύριο 11 με 12.30 και η παρουσίαση του γράφου εργασίας της κυρίας Γκέπαρτ που πρόσβασε ένα βασικό λογαριασμό πληρωμών ε, θα γίνει αύριο. Η έκθεση Πέρες θα είναι την ε, Τετάρτη και από ό,τι φαίνεται την Τετάρτη θα τελειώσουμε στις 16 ε, και 15 αλλά αργότερα. έχω να συναντηθώ για τις δημόσιες προμήθειες με τον Βρετανό Υπουργό. Είναι πρώτη του επίσκεψη για αυτό το θέμα και θα εκπροσωπήσω και την Επιτροπή μας σε μια συνάντηση του Steering Group του διαλόγου για τα διατλαντικά και με το Συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα. Είναι πολύ σημαντικό να έχει λόγο η Επιτροπή μας για τα εμπορικά ζητήματα. Συνεπώς, θα πω το εξής. Έχουμε εδώ πέρα και την κυρία Κόρχολα και την κυρία Βανιό, τους δύο εξέχουσες αντιπροέδρου μας, που θα αναλάβουν. Ε, θα ξανάρθω για να υποδεχτώ τον Επίτροπο Μπαρνιέ, αλλά μετά θα ξαναφύγω. Λοιπόν, εσείς έχετε και ερωτήσεις για τον κύριο Μπαρνιέ. Ωραία, η Μπερναδέτ θα το φροντίσει. Αυτά για σήμερα το απόγευμα. Οπότε συνεχίζουμε και περνάμε ευθύ αμέσω στην ψηφοφορία της έκθεσης της κυρίας Φόξ για την πολιτική ανταγωνισμού. Και μετά θα πάει στην αρμόδια περιουσία επιτροπή ο κύριος Φόξ, ο κύριος Φόξ για να την παρουσιάσει και εκεί. Κύριε Φόξ, τι έχετε να μας πείτε. Το μόνο που έχω να πω, Πρόεδρε, είναι ευχαριστώ πολύ τους και εισηγητές για την βοήθειά τους που δέχτηκαν τους συμβασμούς. Ο κύριος Σβάπ θα λάβει υπόψη του την γνωμοδότηση αυτή όταν ετοιμάσει τη δικιά του έκθεση στην Επιτροπή την Οικονομική. Αυτά, Πρόεδρε, δεν έχω άλλες παρατηρήσεις. Πρόεδρος. Ναι, υπήρχαν διάφορα σημεία. Ε, θα δώσω το λόγο σε όσους θέλουν όσο προχωράμε. Όποιος έχει κάτι να πει, ας κουνήσει το χέρι του να τον δω. Αλλιώς μπορούμε να ξεκινήσουμε με την ψηφοφορία και δεν χρειαζόμαστε τις κάρτες μας, έτσι. Παράγραφος 1, παράγραφος, τροπολογία 1 υπέρ, κατά, α, εγκρίνεται. Τροπολογία 2 μπουζόι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία τώρα στην τροπολογία 3. Ο κύριος ε, Σβάπ νομίζω είχε κάνει κάποιες μικρές αλλαγές στο κείμενο. Σωστά. Θέλετε να μας το διαβάσετε. Πρόεδρε, προσπαθήσαμε, αλλά υπήρχε ένα θέμα διατύπωσης. Λοιπόν, λέει ότι αναμένει προσαρμογή των καθημερινών γραμμών, όπως και του κανονισμού σχετικά με τις επιχειρήσεις ενό προϊόντος και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Αλμούνια. Ωραία. Υπέρ παρακαλώ, λέει ο Πρόεδρος. 13 in favor. Those against. Κατά. Κατά. Εγκρίνεται. Η τρία καταπίπτει Πέντε τώρα του κύριου Πάξας. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Απορρίπτεται σαφέστατα. Τέσσερα. κανθά. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 7. Λουίς Γκρέχ υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τώρα έχουμε συμβαστική τροπολογία αριθμός 1. Αλλά ε, κυρία Χρυσαπίλτ και κύριο Σφάλ πιστεύουν ότι η δικιά τους τροπολογία 30 δεν έχει συμπεριληφθεί στο συμβιβασμό. Οπότε τι θέλουν, θέλουν κάποια αλλαγή. Προτείνω να ψηφίσουμε το συμβασμό πρώτον ως έχει και μετά να δούμε αν θα δεχτείτε να προσθέσουμε και την τροπολογία 30 εκεί. Λοιπόν, συμβαστική αριθμός 1. Υπέρ παρακαλώ. Όχι, δεν είναι σαφές. Μια στιγμή, συγγνώμη, λέει κυρία Γεπάρτ. Είμαι σκιώδη συζήτρια της ομάδας μου και εγώ δεν ξέρω για ποια προσθήκη μιλάτε. Οπότε λυπάμαι, δεν μπορώ να αποφανθώ για τέτοια προσθήκη. Δεν την ξέρω.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 Λοιπόν, θα ψηφίσουμε πρώτα το συμβασμό. Ψηφίζουμε τη συμβαστική τροπολογία αριθμό 1, παρακαλώ. Γιατί έτσι καλώ πρέπει να το ψηφίσουμε. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τώρα το ερώτημα είναι. Και τι προτείνω. Προτείνω να ψηφίσουμε την τροπολογία 13 ως προσθήκη και θα δείξει αν συμφωνείτε ή όχι. Νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε. Εντάξει. Τροπολογία 13, ε, ως έχει. Και πρόκειται για τα συμπληρώματα διατροφής που λέτε ότι δεν καλύπτεται. Συγγνώμη, λέει η κυρία Κέπχαρτ, λυπάμαι, αλλά τέτοιου είδου πράγματα πρέπει κανεί να τα λέει από πριν. Και όχι έτσι ξαφνικά να παρουσιάζει κανείς ένα κατάλογο ψηφοφορίας τέτοιων. Και μετά να τον αλλάζουμε στην ψηφοφορία. Δεν ε, πρέπει να γίνονται αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό και θεωρώ πως αυτή η διαδικασία είναι αντίθετη με τον κανονισμό μας ανεξαρτήτως του πόσο καλή μπορεί να είναι αυτή η τροπολογία 13. I mean, I have... Πρόεδρος, δεν θέλω να χάσουμε χρόνο τώρα το συμπαθούμε. Εντάξει, κατανοώ αυτό που λέει η κυρία Κέπαρ. Δεν νομίζω ότι είναι και τόσο σημαντικό. Νομίζω ότι είχε συζητηθεί με του Σκιώδη. Εφόσον δεν συζητήθηκε και δεν συμφωνήθηκε με του Σκιώδη, νομίζω και εγώ ότι δεν είναι σωστό να το βάλω σε ψηφοφορία εδώ σε αυτή τη συνεδρίαση. Αν θέλετε λοιπόν αυτά τα σημεία να τα προσθέσετε αργότερα, έχετε την ευκαιρία στην Ολομέλεια να το κάνετε αυτό. Εξάλλου, μια γνωμοδότηση είναι αυτή που κάνουμε στην Οικονομική Επιτροπή, έτσι. Αυτά. Και η κυρία Κέπαρ νομίζω ότι έχει δίκιο νόμιζα ότι είχε συζητηθεί με τους σκιώδες προηγουμένως. Εάν όμως μία ομάδα δεν συμφωνεί, τότε πρέπει να το δεχτείτε αυτό. Σίγουρα ένα στοιχείο της 13 συμπεριλαμβάνεται στο συμβασμό που μόλις εγκρίναμε. Άρα νομίζω ότι συγκεκριτής έτσι κι αλλιώς είναι... Ε, έχει κάνει περισσότερο από πολλά. Όχι, όχι, δεν θέλω να το συζητήσουμε. Ζητάει το λόγο κυρία Κορέτσα. Δεν την ακούμε. Μιλάει εκτός μικροφώνου. Ωραία, έχετε το λόγο, κυρία Κοράτσα. Τι διαδικαστικό έχετε, θα μου θυμίσετε, θα μου λύσετε επί του κανονισμού, έτσι, όχι επί του περιεχομένου. Έχω δικαίωμα να ζητήσω η τροπολογία μου να ψηφιστεί ε, ο κύριο Σφάλτ και εγώ πιστεύουμε ότι δεν συμπεριλαμβάνεται. Σήμερα στι 11.30 πήραμε το κατάλογο ψηφοφορία. Ερχόμαστε από τη Στοκχόλμη. 2 ώρε και 45 λεπτά ταξίδι. Πήρα ένα SMS όταν έφτασα στο αεροδρόμιο. Ε, συγγνώμη, το πρόβλημα είναι ότι πήραμε πάρα πολύ αργά τον κατάλογο ψηφοφορία. Αλλά δεν μπορείτε εσεί να τα βάζετε μαζί μα και να λέτε ότι έπρεπε να το έχουμε κάνει νωρίτερα. Δεν είχαμε χρόνο, ήταν αδύνατον να κάνουμε οτιδήποτε πιο πριν. Στι 3 εγώ βλέπω το κείμενο. Έφτασε όλοι καθόντουσαν ήδη εδώ. Υπάρχει ένα διαδικαστικό ζήτημα εδώ, Πρόεδρε. Και δεν είναι ότι εμεί αργήσαμε, είναι ότι ο κατάλογο ψηφοφορία έφτασε αργά. Εμεί δεν θεωρούμε ότι η τροπολογία αυτή 13 αποτελεί μέρο τη συμβαστική. Ήταν δικιά μου έκθεση για μια πιο δίκαια λιανική αγορά στην Ευρώπη και νομίζω ότι έχω δικαίωμα να μιλήσω γι' αυτό. Και αν δεν υπάρχει πρόβλημα επί της ουσίας, θα ήθελα οι συνάδελφοι να το σκεφτούν είναι θέμα διαδικαστικό. Εξαιτία διαδικασία δεν μπορούσα να το είχα κάνει νωρίτερα. Και δεν, υπάρχει, δεν είναι επίμαχο, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανεί που διαφωνεί. Παρακαλώ τη 13α λοιπόν να την ψηφίσουμε χωριστά εκτό του σεβασμού. Και ειλικρινά θα ήμουν ευγνώμων προ του συναδέλφου αν δεχτούν να το κάνουμε αυτό. Πρόεδρο, η γραμματεία μου λέει ότι την Παρασκευή το απόγευμα ήταν έτοιμο κατάλογος ψηφοφορία. Οπότε, αν το είδατε εσεί ή όχι τότε, αυτό είναι άλλο θέμα. Για να δούμε λοιπόν. Όλα θα εξαρτηθούν από τη στάση και των υπόλοιπων πολιτικών ομάδων. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα περισσότερο. Όπως και να έχει το πράγμα πάντως. Μέρος της τροπολογίας στις 13 συμπεριλαμβάνεται πρώτα απ' όλα ε, στο συμβασμό. Από ό,τι καταλαβαίνω θέλετε και ένα άλλο κομματάκι της δικιάς σας τροπολογίας που δεν συμπεριλαμβάνεται και θέλετε αυτό να προσθεθεί στην ε, συμβιβαστική. Για να δούμε. Ας προσπαθήσω να το διαβάσω και να δούμε αν ε, υπάρχει κανείς που έχει... Α, αντίρρηση. Α, θα έχετε σαν αντίρρηση. Ε, τότε δεν έχει νόημα να το κάνω. Η κυρία Γκέπχαρτ. Ναι, μα το θέμα δεν είναι το περιεχόμενο, αλλά η διαδικασία. Δεν επιτρέπεται αυτή η διαδικασία. Διαπιστώνω δε, ειδικά από το ΕΛΚ τελευταία, πως γίνονται συμβαστικές τροπολογίες και μετά ξαφνικά έρχονται χωριστές ε, τροπολογίες ή προφορικές τροπολογίες ε, που κατατίθενται εκ των υστέρων. Ε, δεν είναι αυτή η αξιοπιστία για να δουλέψουμε. Γι' αυτό και δεν το δέχομαι. Έχουμε τη δυνατότητα να το ξαναδούμε το θέμα στην Επιτροπή, στην Ολομέλεια και εκεί να καταθέσουμε τροπολογίες. Αλλά σήμερα δεν δέχομαι να ξανανοίξουμε το συμβιβασμό που είχαμε επιτύχει και να ξαναρχίσουμε να το συζητάμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Well, I mean, on basis, that βάσεις φοβούμαι πως δεν θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε και θα πρέπει να το ξανακαταθέσετε. Να το δώσετε στον κύριο Φόξ και να προσπαθήσετε να περάσει στην Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή. Τώρα, εγώ από ό,τι κατάλαβα η συμβαστική είχε συμφωνηθεί από το ΕΛΚΑ την περασμένη εβδομάδα, την Πέμπτη μάλιστα. Λυπάμαι αν δεν ε, θεωρείτε ότι δεν είχατε αρκετό χρόνο, αλλά η γραμματεία ακολούθησε τη σωστή διαδικασία πάντως. Ας προχωρήσουμε. Now on amendment 14. Πάμε στην ε, τροπολογία 14 Γκέπχαρτ, όπου έχει ζητηθεί κατά τμήματα ψηφοφορία από την ΕΣΥΑΡ, το έχετε στα εγγραφά σας. Τμήμα 1 ψηφίζουμε, ποιοι είναι υπέρ. Το ΕΛΚ ψηφίζει από αυτού. Τι θα κάνετε απεργία? Είστε ένδειξη μαρτυρίας? Όχι. Λοιπόν, υπέρ κατά, ε, εγκρίνεται το πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα, ποιοι είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στην τροπολογία 15, Γκέπχαρτ, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Συγγνώμη, πρέπει να μετρήσουμε. Υπέρ ποιοι είναι. Those Κατά. Καταπίπτει γιατί είχαμε σοπαλία. 21, υπέρ. Uh, Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Συμβαστική υπέρ, κατά. Ποχές. εγκρίνεται. Και φτάνουμε στην 24. Καμφά, υπέρ, απορρίπτεται. Συμβαστική τρία υπέρ κατά αποχές γίνεται. Τροπολογία διαγραφής 25 του κυρίου Σαλβίνη υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 26 Μπουζόη υπέρ. Πρέπει να μετρήσω. Ποιοι είναι υπέρ της 26.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 Τροπολογία 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ κατά απορρίπτεται. 31 υπέρ, ως προσθήκη υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ, Κατά. Ναι, εγκρίνεται. 33 καμφά Κατά. Απορρίπτεται. 35 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 36 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 37 έχει ζητηθεί ψηφοφορία κατά τμήματα από την ΕΣΥΑΡ Τμήμα 1 Ποιοι είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τμήμα 2, υπέρ. Those against. Κατά. Those against. Were you voting in favour, Mrs. Le Grip, were you? That, so that's rejected. Απορρίπτεται, 11-11. 38 καμφά υπέρ κατά απορρίπτεται. Και περνάμε τώρα στην τελική ψηφοφορία για το σχέδιο γνωμοδότησης. Ποιο είναι υπέρ. Uh, so that's okay. Those in favour, you can count the numbers. No, you don't need to count because we'll see who's against and subtract. So we haven't. Those against, abstention κατά αποχές εγκρίνεται 21 21 ψήφι καμία κατά, καμία αποχή. Σας ευχαριστούμε πολύ και θα προσπαθήσουμε να στηρίξουμε αυτή τη γνωμοδότηση στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων. Κύριος Σβάμπ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως δεχόμαστε την απόφαση, συγχαίρουμε τον κύριο Φόξ. Να σας πω μόνο πως αύριο η σοσιαλιστική ομάδα που δεν θέλει και αυτή να είναι αναξιόπιστη επίσης ε, θα ζητήσει ε, προφορική ψηφοφορία Οπότε και εμείς, η κυρία Γκέπχαρτ αύριο, τροπολογίες ε, των ε, σοσιαλδημοκρατών που θα έρθουν ε, αργά, θα είμαστε αναγκασμένοι να τις καταψηφίσουμε. Παρόλο που και εμείς μπορούμε να συμφωνούμε. Έτσι θα γίνεται μέχρι να κοιτάει κανείς την ουσία και όχι τη διαδικασία. Ευχαριστώ. Ε, ο Πρόεδρος, δεν θέλω τώρα να διαταράξω το, κλίμα της Επιτροπής... Εύελιν Γρήγορα. Όπως είπατε, αύριο θα υπάρξουν προφορικές τροπολογίες, αλλά όπως έχουμε ήδη πει, βλέπετε πως ήδη εσείς το ξέρετε. Το γνωρίζετε ήδη. Εδώ πέρα όμως, τι συνέβη σήμερα, στη μέση της ψηφοφορίας, χωρίς πληροφόρηση σκιωδών εισηγητών και συντονιστών, ε, συνέβη αυτό. Ε, εδώ πέρα υπάρχει μια μικρή διαφορά ανάμεσα στι δύο περιπτώσεις. Ο πρόεδρος, μάλιστα. Ελπίζω να συνεχιστεί η συνήθι πρακτική και σας υπενθυμίζω προσπαθούμε να μοιράσουμε τον κατάλογο ψηφοφοριών. Οι σύμβουλοι σας θα παρακολουθούν, πρέπει και εσείς να δείχνετε λίγη προσοχή. Τώρα θα αναλάβει την ε, Προεδρία η συνάδελφος και τα λέμε σε λίγο. Okay, good afternoon. We now move uh, Καλησπέρα, προχωράμε. Έχουμε εδώ να κάνουμε με την συμφωνία για τα στεγαστικά δάνεια και δίνω το λόγο στον εισηγητή κύριο Λέχνε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ακίνητα κατοικία. Λοιπόν, είχαμε και μια σύντομη συζήτηση για την έκθεση αυτή με, τον, με τους ηγητές. Έχουμε συμφωνήσει σχεδόν για τις μισές τροπολογίες. Να πω ε, τέλος πως ε, είμαστε κατά της διεύρυνσης του πλαισίου το οποίο έχει προτείνει η Κομισιόν και θέλουμε εμείς περισσότερο να γίνει αυστηρότερο το πλαίσιο γι' αυτό. Ζητήσαμε από τους ε, συναδέλφους να στηρίξουμε την έκθεση της ε, Κομισιόν κάτι με το οποίο εγώ συμφωνώ εγώ στην έκθεσή μου προσπάθησα να ακολουθήσω μία μέση οδό και να υποβάλω μία έκθεση η οποία θα ακολουθεί τη γραμμή ε, που προαναφέραμε βεβαίως υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι που θέλουν να επεκτείνουν κατά πολύ την έκθεση. Όπως ακριβώς έχει γίνει με την έκθεση της Περσέδο στην ΕΚΟΝ. Υπάρχουν κάποια πράγματα με τα οποία μπορούμε να συμφωνήσουμε, με κάποια άλλα όχι. Υπάρχουν κάποια ζητήματα στα οποία έχω αμφιβολίες για το εάν ε, μπορούν να ισχύσουν για ολόκληρη την Ευρώπη και να ξέρουμε ποιες θα είναι οι συνέπειές τους. Δηλαδή, αν το σκέφτεται κανείς στο εθνικό πλαίσιο, και αν ήταν σε μία ε, λευκή βίβλος θα μπορούσα οπωσδήποτε να τα δεχτώ αλλά τώρα χωρίς μελέτες να τα προτείνουμε για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα ήθελα να το κάνω. Αυτό το οποίο μπορεί να ισχύει σε μια χώρα μπορεί να είναι τελείω λανθασμένο για μια άλλη. Να φέρω ένα παράδειγμα. Μια τροπολογία, δεν ξέρω, είναι για πολλέ τροπολογίες. Η 205 στο άρθρο 9α που απαγορεύει την σύνδεση, αν θέλετε. Μια χαρά ιδέα, αλλά να σα υπενθυμίσω πω στη Γερμανία υπάρχει ένα επιχειρηματικό μοντέλο με τζίρο πάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ, στην οποία τα ταμιευτήρια προσφέρουν συνολικά δάνεια πιστώσεων ε, σε συνδυασμό με μια άλλη τράπεζα που δεν είναι ταμιευτήριο. Ακριβώς όλα αυτά προς συμφέρον του καταναλωτή, του μικροκαταναλωτή. Αυτομάτως πλέον αν απαγορεύσουμε τέτοιες διασυνδέσεις θα απαγορευτούν όλα αυτά τα πράγματα και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα. Και με όλα αυτά δεν ξέρω εάν ακολουθούμε το σωστό δρόμο. Επίσης, σε πολλά σημεία τα οποία εντάξει μπορεί να έχουν καλή πρόθεση το εάν μπορούν να ισχύσουν όμως σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ή αν θα μπορούσαν ίσως τα προβλήματα αυτά να αντιμετωπιστούν με εθνική αντιμετώπιση νομίζω θα ήταν καλύτερο αυτό. Τέλος, δεν συμφωνώ με κάποιες άλλες προτάσεις όχι γιατί είναι λάθος, αλλά δεν είναι συνεπής με την νομοθεσία συνολικά. Είχα πει και στην πρώτη μου τοποθέτηση και επιμένω σε αυτό πως θα πρέπει να προσπαθήσουμε όταν μιλάμε για τον ίδιο τομέα να μην αποκλίνουμε. Δεν μπορούμε να λέμε στα κράτη-μέλη και στους ανθρώπους για την ίδια περίπτωση πως υπάρχουν δύο διαφορετικές ε, νομοθεσίες και ο Ευρωπαίος νομοθέτης καμιά φορά πρέπει να σκέφτεται τι ε, στέλνει στον εθνικό νομοθέτη για να ληφθεί και το ζήτημα επίσης να διευκολυνθεί και το ζήτημα της μεταφοράς. Επίσης, είναι άλλη η καταναλωτική πίστη από τα στεγαστικά δάνεια. Αλλά δεν ξέρω τώρα με τη διατύπωση τι θα γίνει. Ομολογώ επίση πω πάρα πολλοί συνάδελφοι είναι υπέρ τη διαγραφή πολλών πράξεων κατά εξοδότηση. Τώρα, για το θέμα της Επιτροπής ε, Οικονομικών. Πράγματι δεν μπορούμε να δούμε το θέμα αυτό μόνο υπό το πρίσμα της προστασίας των καταναλωτών, αλλά και υπό το πρίσμα της ε, χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Οπότε πράγματι και η Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων έχει εδώ πέρα άποψη. Αλλά δεν θα πρέπει να έχουν την πλήρη και αποκλειστική αρμοδιότητα για την πρόταση αυτή. Να αφαιρθώ σε κάποια πράγματα συγκεκριμένα πεδίο εφαρμογής. Εδώ, συνάδελφος Φόξ, κυρία Κοχόλα και άλλοι έχουν προτείνει ένα περιορισμό. Εν μέρη συμφωνώ. Αλλά από την άλλη κάπου παραπάει. Σύμφωνα με την πρόταση δηλαδή του κυρίου Φόξ θα μιλάμε μόνο για κίνητα τα οποία χρησιμοποιεί ο ίδιος ο αγοραστής. Ε, αυτό παραπάει. Δηλαδή χάνεται το νόημα με τα χρηματοπιστωτική σταθερότητα κτλ. Αλλά υπάρχει μια τροπολογία που λέει κανένα δάνειο πάνω από 2 εκατομμύρια. Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ εκτεταμένη η οδηγία αυτή και ε, ξέρετε πως η κατάσταση διαφέρει από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. Μιλάμε πράγματι για ε, κίνητα κατοικίας και η οδηγία καλύπτει ε, οποιοδήποτε ακίνητο το οποίο αγοράζει με δάνειο, ακόμα και αν είναι επαγγελματική στέγη. Τώρα δεν ξέρω εάν ε, πέντε τραπεζίτες που να χτίσουν ένα εργοστάσιο. Δεν ξέρω αν έχει νόημα να υπαχθεί το... η περίπτωση αυτή στην οδηγία μας. Τώρα. Άλλος συνάδελφος είπε σε κάθε πτυχή να έχουμε την ελάχιστη εναρμόνιση. Εγώ θα πρότεινα στις ε, επεξηγήσεις ε, να το αναφέρουμε. Να αναφέρει δηλαδή η Κομισιόν πως δεν έχουμε εξαντλήσει τα πάντα. Αλλά ορισμένα πράγματα είναι αποφασιστικά. Πρέπει να το πει αυτό η Κομισιόν. Δηλαδή το ετήσιο πραγματικό επιτόκιο. Η... Ε, για μένα είναι ξεκάθαρο ούτω ή άλλω. Ε, προκύπτει από το κείμενο ότι πρόκειται για ελάχιστη εναρμόνιση. Ε, ορισμένα πράγματα μόνο πράγματα εναρμονίζονται πλήρω. Επίσης δεν θέλω να εισαχθούν ε, καινούργιοι ορισμοί και θα πρέπει να τηρήσουμε νομίζω την οδηγία περί καταναλωτικής πίστης. Τώρα, ο αξιολογητής, αυτό που λέγεται αξιολογητής ακινήτων είναι πολύ πολύ πολύ πολλοκός ορισμός. Εγώ δεν ξέρω αν έχει κάνει κάποιο νόημα. Δηλαδή θα πρέπει οπωσδήποτε για κάθε δάνειο να υπάρξει κάποιος ανεξάρτητος δε ο οποίος θα κάνει την ε, εκτίμηση ε, ακριβένουμε έτσι το, το δάνειο την πίστη δεν, δεν έχει νόημα ας τα αφήσουμε νομίζω στον ανταγωνισμό τελευθούμε από το ευρωπαϊκό επίπεδο και να πούμε αναγκαστικά για κάθε ενυπόθηκο δάνειο θα πρέπει να υπάρξει αξιολόγηση μέσω μιας άλλης επιπλέον αρχής, ε, η υπηρεσία ή οτιδήποτε, θα, θα ακριβίνει έτσι η πίστη. Δεν είναι δυνατόν. Θα πρέπει σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Και δεν είναι και προς το συμφέρον του καταναλωτή, όπως είπα, γιατί κοστίζει. Για τις αρχές. Να πω πως εγώ είμαι κατά του να έχουμε συνεχώς νέες αρχές και υπηρεσίες. Έχουμε αρκετές. Στο άρθρο 5 προς το συμφέρον του καταναλωτή προτείνουμε εδώ πέρα πως πράγματι η δραστηριότητα των υπαλλήλων της τράπεζας θα ε, πρέπει να είναι επαγγελματική. Αλλά το να λέμε τώρα προς το συμφέρον του καταναλωτή, ε, είναι προς το συμφέρον της τράπεζας, να κάνουμε. Ε, δηλαδή θα, θα πάει προς την αντίστοιχη πλευρά. Τώρα, διαφήμιση ο κύριος Μπούζε, δεν ξέρω τι εννοεί εδώ πέρα. Θα μπορούσα, εν πάση περιπτώσει, να συμφωνήσω σε κάποιες συντομεύσεις για να μην το παραφορτώσουμε για τη διαφήμιση. Το άρθρο 9 τώρα δικαίωμα υπαναχώρησης. Για το δικαίωμα αυτό λοιπόν υπαναχώρηση για τις τυποποιημένε πληροφορίε. θα πρέπει να έχει το χρόνο να σκεφτεί την απόφασή του βεβαίω. να δούμε αν θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια συμβαστική λύση. Η απαγόρευση, όπως σας είπα, διασυνδέσεων συνεργασιών, είπα ήδη κάποια πράγματα, ετήσιο πραγματικό επιτόκιο. Νομίζω πως σωστό είναι αυτό το οποίο έχουμε προτείνει και ήδη άρθρο 14, η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας, ε, λέει θα πρέπει πράγματι να ε, λαμβάνεται υπόψη και να είναι κάπως ε, συγκρίσιμη με την οδηγία περί καταναλωτικής πίστης. Το αρθρο D14 και η Κομισιόν έχει πει πως είναι κάτι το σημαντικό, πως εάν είναι αρνητική η αξιολόγηση αυτή δεν ε, μπορεί να υπάρξει κάποια εγγύηση του δανείου. Εδώ πέρα απαγορεύουμε ουσιαστικά μια εμπορική συναλλαγή. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Γιατί υπάρχει ούτως ή άλλως. Ξέρετε πως και αυτές οι αξιολογήσεις είναι προβληματικές. Και τι θα οδηγήσουμε εδώ πέρα σε ένα σύστημα στο οποίο δεν θα δίνονται καθόλου δάνεια. Οπότε θεωρώ εγώ είτε να το διαγράψουμε αυτό το οποίο ζήτησαν αρκετοί συνάδελφοι, είτε όπως εγώ ζήτησα να το αναδιατυπώσουμε για να έχει την έννοια της εποπτείας. Δηλαδή ε, να πρέπει να δικαιολογηθεί ε, το πιστοτικό ίδρυμα έναντι της ε, εποπτεύουσας αρχής, αλλά να μην έχει την έννοια του δικαίου για να απαγορεύει μια σύμβαση. Τέλος για το άρθρο 18. Εδώ πέρα πολλοί συνάδελφοι και εγώ έχουν κάνει αρκετές διορθώσεις. Πρέπει να υπενθυμίσουμε πως διαφέρουν πάρα πολλοί καταστάσεις στα κράτη-μέλη. Στη Γερμανία πάνω από 80% των στεγαστικών δανείων ε, δίνονται με σταθερό δάνειο, με σταθερό επιτόκιο, με συγχωρείτε, Επίσης και το θέμα της ε, ποινή ε, προεξόφλησης ε, έχει ρυθμιστεί από πάγια νομολογία. Αυτό το οποίο θα έπρεπε να σκεφτούμε είναι αυτό το οποίο προτείνει ο κύριος Γκοκ, νομίζω. Αν έχουμε δηλαδή μια προεξόφληση του δανείου, αυτό μήπως είναι και πλεονέκτημα για την τράπεζα. Μήπως δηλαδή θα έπρεπε και να αποζημιωθεί ο δανειολήπτης. Μήπως αυτό να σκεφτούμε. Το, το, μηδέν, το, μηδέν είναι ισχύει ούτως ή άλλως ε, κύριε συνάδελφε. Αλλά εάν επωφελείται και η τράπεζα, δεν ξέρω, θα πρέπει να το δούμε και αυτό. Όπως σας είπα έχουμε το 18α, τώρα για την ε, αξιολόγηση αυτή δεν θα είμαι υπέρ. Τέλος, για το χρονοδιάγραμμα. Δεν ξέρω οι συνάδελφοι ε, τι άποψη έχουν. Δεν, δεν ανάγκη νομίζω να ισχύσει για έξι χρόνια όπως για την οδηγία καταναλωτικής πιστής, αλλά εάν είχαμε μείνει στο πλαίσιο της ε, Κομισιόν και σε πέντε χρόνια κάνουμε το επόμενο βήμα, νομίζω πως ε, θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία εγκαίρως. Αλλά θεωρώ πως ε, αποκλείεται θέματα τα οποία είναι ευθύνη και δική μα και τη Επιτροπή Οικονομικών να μην ολοκληρωθούν μέχρι το τέλο του έτου. Οι σκιώδει ηγητέ ε, θεωρούσαν ομόφωνα πω στι 5 Δεκεμβρίου δεν πρέπει να ψηφίσουμε, αλλά πως χρειάζεται λίγο χρόνο παραπάνω για να σκεφτούμε το ζήτημα. Γιατί η ΕΚΟΝ λέει γιατί δεν το ξέρω εγώ κτλ. δεν ξέρω γιατί βιαζόμαστε, θα πρέπει το Κοινοβούλιο να ενημερωθεί επαρκώ. Αλλά αυτό σημαίνει πως και εμείς ε, δεν νομίζω να πρέπει να ψηφίσουμε στις 5 με Αυτά κυρία Πρόεδρε. Um, Σα ευχαριστώ. Πρέπει να σας ειδοποιήσω ότι πρέπει να είμαστε ακριβείς. Όταν έρθει ο κ. Μπαρνιέ, πρέπει να είμαστε στην ώρα μας για να μπορέσουμε να τον ακούσουμε. Αυτό που θα κάνουμε είναι να δώσουμε το λόγο στους και ηγητές όσο επιτρέπει ο χρόνος και... και μετά θα αρχίσουμε στην ώρα μας. Ξεκινάμε με τον κύριο Χουάνγκ Γκόγκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Λέχνερ για το σχέδιο χρηματοδότησης γιατί το θέμα αυτό είναι εξαιρετικά ευαίσθητο και λεπτό και παρά στην, τη λεπτομερή του παρουσίαση ομολογώ ότι κάπως έχω απογοητευτεί από τις προτάσεις του. Βέβαια καταλαβαίνω ότι πρέπει να μείνουμε μέσα στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Επιτροπής μας και να μην μπούμε στα νερά άλλης Επιτροπής, αλλά δεν μπορούμε να αρκεστούμε στο να ευθυγραμμίσουμε αυτήν την οδηγία στην οδηγία ε, για την ε, καταναλωτική πίστη. Εφόσον μιλάμε για στεγαστικά δάνεια ε, και τα συζητούμε χωριστά, αυτό γίνεται γιατί δεν μπορούν να αξιομοιωθούν με τα καταναλωτικά. Για δύο λόγους. Καταρχήν, γιατί η διάρκεια των καταναλωτικών δανείων είναι σημαντική. Όχι, διορθώνει ο μιλητής. Ενώ τα καταναλωτικά δεν είναι σχετικά σύντομες περίοδοι. Ε, τα στεγαστικά δεσμεύουν τον καταναλωτή για 15, 20, 25 χρόνια της ζωής του. Δεύτερον, ο συστημικός κίνδυνος μέσω αυτών των στεγαστικών δανείων ε, για τα οποία η κρίση των subprime ήταν ε, φατρανή απόδειξη, οδηγούν σε, μας κάνουν να κατανοήσουμε ότι είναι ιδιαίτερη φύση αυτών των δανείων. Εμεί στην ομάδα μου θεωρούμε ότι Αυτά τα στεγαστικά δάνεια θα πρέπει να είναι αντικείμενο κανόνων που θα λαμβάνουν υπόψη στι ιδιαιτερότητε, θα προστατεύουν καλύτερα ε, κατά των καταχρηστικών ε, πρακτικών του καταναλωτέ, θα προλαμβάνουν την αδυναμία ε, αποπληρωμή, χωρί να εμποδίζουν όμω του πιο χαμηλόμιστου καταναλωτές να μπορούν και αυτοί να έχουν δάνεια. Το σχέδιο χρηματοδότηση είναι ιδιαίτερα διστακτικό κατά τη γνώμη μας. Κάποιες πρακτικές θα πρέπει να σταματήσουν γιατί αποτελούν κατάχρηση από πλευρά των πιστωτών απέναντι στους καταναλωτές οι οποίοι είναι λάθος. Δηλαδή, επιβάλλουν στους καταναλωτές που θέλουν πιο γρήγορα να αποπληρώσουν το δάνειό τους τέτοιου είδους ποινές ε, και οικονομικές κυρώσεις που δεν ε, τους συμφέρουν να το κάνουν. Επίσης, το να δώσει κανείς ε, την έγκρισή του δεν πρέπει να υποχρεώνει τον καταναλωτή να κάνει ασφαλιστικό συμβόλαιο στην ίδια τράπεζα. Ο καταναλωτής θα πρέπει να μπορεί να κάνει την ασφάλισή του εκεί όπου επιλέγει. Χωρίς αυτό να επηρεάζει την προσφορά την δανειακή που του γίνεται. Ε, ορίστε παραδείγματα συγκεκριμένων κανόνων που θα ήθελα να περιλαμβάνονται σε αυτό το κείμενο της οδηγίας γιατί έτσι <coughs> θα μπορέσει να αποκατασταθεί η σχέση ανάμεσα στους δανειοδότες και τους καταναλωτές. Ναι, ναι, ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος. Ο κ. Μπουσουτήλ έφυγε πολλά από αυτά τα οποία είπε ο κύριος Λέχνερ. Ναι, επί της αρχής μας βρίσκουν σύμφωνος και θα έπρεπε νομίζω να αναβληθεί η ψηφοφορία επί της έκθεσης για να μπορέσουμε να έχουμε και περισσότερες ε, συμβαστικές τοπολογίες. Ευχαριστώ. Okay, thank you. Ευχαριστώ κυρία Ρούλε. Μια στιγμούλα, ναι. Ευχαριστώ στους και οδησίγητες. Υποστηρίζω την πρόταση να προσπαθήσουμε να μην ψηφίσουμε 5 Δεκεμβρίου, γιατί δηλαδή λόγω των πολλών τροπολογιών πρέπει να δούμε μήπως μπορούμε να έχουμε συμβιβαστικές τροπολογίες. Και τέλος, να πω πως εγώ ήμουν επιφυλακτική εξ αρχής απέναντι σε αυτήν την τροπολογία λόγω των προβλημάτων που είχαμε σε κάποια κράτη-μέλη με τα στεγαστικά δανεία. Θεωρώ ιδιαίτερα προβληματικό γιατί έχουμε, το έχουμε διαπιστώσει αυτό και στην Πράσινη Βίβλο πως υπάρχουν μεγάλες διαφορές στα κράτη-μέλη πως οι καταναλωτές έχουν διαφορετικές κουλτούρες όσον αφορά τα ενυπόθηκα δάνεια και δεν έχει νόημα να έχουμε ε, πανευρωπαϊκές ρυθμίσεις. Θεωρώ πως θα πρέπει να μείνουμε στην ελάχιστη εναρμόνιση. Επίσης θεωρώ πως και οι πράξεις κατεξοδότηση πρέπει να διαγραφούν στο μέτρο του δυνατού και να τονίσω πως υπάρχουν ελάχιστες διασυνοριακές ε, ε, πιστώσεις ενυπόθηκες και άρα δεν θεωρώ πως πρέπει να υπάρξει κάποια ευρωπαϊκή ρύθμιση. Πρέπει να έχουμε τις βασικές αρχές προστασίας των καταναλωτών και τέλος. Σε πέντε χρόνια ίσως μπορούμε να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα. Ε, επίσης θεωρώ πως θα πρέπει να υποβληθεί μια μελέτη επιπτώσεων για ορισμένα πράγματα γιατί δεν μπορούμε να κρίνουμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις σε κάποια κράτη-μέλη και δεν είναι λογικό να πηγαίνουμε στο άγνωστο. Mr. Fox, Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή για τη δουλειά που συνεχίζει να κάνει για αυτό το θέμα. Συμφωνώ με την κυρία Ρούλε για το ότι υπήρξε πραγματικά πλήρης έλλειψη ε, δεν λάβαμε δηλαδή, καθόλου υπόψη μας στο διασυνοριακό εμπόριο σε αυτή την περίπτωση και συμφωνώ με αυτά που είπε για τις κατεξοδότηση πράξεις. Ο κύριος Λέκνερ γνωρίζει τις απόψεις μου όσον αφορά τις υποθήκες ότι θα έπρεπε να βγουν από την οδηγία αυτή. Εγώ είπα ότι είναι εμπορικές οι υποθήκες αυτές. Και γι' αυτό, κατά τη γνώμη μου, για μένα δεν πρέπει να εμπίπτουν ε, στα πλαίσια της οδηγίας αυτής. Και κάτι παραπάνω που θέλω να πω είναι το εξή Αυτό το ίσες που είναι το φυλάδιο αυτό το ενημερωτικό, το ευρωπαϊκό που απαιτούμε, το ίσες. Να ξέρετε ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο έτσι κι αλλιώς υπάρχει ήδη ένα στάνταρ τέτοιο έντυπο το οποίο δίνει τις πληροφορίες που θέλουμε. Το να είναι τώρα ευρωπαϊκό δεν πρόκειται να βοηθήσει τίποτα παραπάνω, θα επιβάλλει παραπάνω κόστος. Οπότε ρωτάω τους ε, συναδέφους, για ποιον το κάνουμε. Το κάνουμε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να μπορεί να πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ορίστε, τυποποίησαμε άλλο ένα έντυπο. Είναι για τους ε, ε, Βρετανούς καταναλωτές. Γιατί δεν είναι σίγουρα για κανέναν άλλον. Και να ξέρετε ότι το ίδιο πράγμα το συζητάμε και για τις άλλες χώρες. Το να υπάρχει ένα τέτοιο έντυπο τυποποιημένο που να μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι διάφορες χώρες είναι έχουν ένα δικό τους. Ο βασικός μας στόχος έτσι κι πρέπει να είναι η προστασία του καταναλωτή και όχι η τυποποίηση για την τυποποίηση. Κάποιο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλό θα κάνει να βρει κάτι άλλο αν θέλει να αισθάνεται καλύτερα. Τώρα συμφωνώ για τι απόψει του κύριου Λέκνερ Επίση ότι δεν πρέπει να πιεστούμε για το Δεκέμβριο. Εγώ δεν ξέρω γιατί η, Οικονομική Επιτροπή βιάζεται τόσο πολύ. Κύριε Λέκνερ, νομίζω ότι ακούσατε ομόφωνα οι σκιώδει οι σα στηρίζουν. Ευχαριστώ. Άλλο κανεί θέλει το λόγο, λέει πρόεδρο. Υπάρχει κάποιο άλλο ευρωβουλευτή που θέλει το λόγο. Όχι. Τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακαλώ η Τζένιφερ Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη και εγώ, γιατί θα έρθει και ο πίτροπος όπου να είναι. Έχω μερικές παρατηρήσεις. Ναι, θα προσπαθήσω να μην επαναλάβω τα σχόλια του Φίλιπ Δελ την προηγούμενη φορά που ήταν εδώ. Νομίζω ότι εξήγησε αρκετά ξεκάθαρα γιατί θέλουμε να συνάδουμε με την οδηγία για τις υποθήκες και σε αυτόν και σε κάποιους άλλους τομείς. Αλλά θέλω να πω δύο λόγια τώρα για κάτι άλλο. Όσον αφορά τις υποθήκες και τις σχετικές συμβάσεις, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε θετικά ίσως κάπως τις τροπολογίες οι οποίες ε, απαγορεύουν ε, το εύρο να συμπεριληφθούν και άλλα οικονομικά προϊόντα και να μπορούμε να προβλέψουμε και κάποιες εξαιρεσει για ορισμένα προϊόντα, για ορισμένου τομείς. Θα δούμε ποια θα είναι η τελική διατύπωση πάνω στην οποία θα συμφωνήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όσον αφορά τώρα το επίπεδο εναρμόνισης, νομίζω ότι εμεί έχουμε προτείνει κάτι πολύ ισορροπημένο. Ανώτατη εναρμόνιση σε ορισμένου τομείς, όπω το EPRC, όπου θέλουμε να κρατήσουμε τους αρχικούς ε, ορισμούς. Συγχρόνως όμως πολλές από τις ε, διατάξεις ε, μιλάνε για εναρμόνιση επί της αρχής. Πράγμα που σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη στην περίπτωση αυτή έχουν μεγάλη ελαστικότητα για να εφαρμόσουν όπως νομίζουν καλύτερα το μέτρο. Γι' αυτό και πιστεύω ότι είναι καλά ζυγισμένη η πρόταση. Αυτά είναι τα δύο κύρια σημεία στα οποία ήθελα να αναφερθώ. Ο κύριος Φόξ θέλει να πω κάτι για το ίσως. Ναι, η SOS. Πιστεύουμε ότι πρέπει η μορφή του εντύπου αυτού να είναι όσο γίνεται πιο εναρμονισμένη. Τώρα, οι κατευθυντήριες γραμμές για την ε, ε, συμπλήρωση του εντύπου να επιτρέπει περιθώρια λιγμού και θα, από αυτού θα έχουμε μια ελάχιστη εναρμόνιση. Έχουμε κάνει μια έκθεση αντικτύπου ανεξάρτητη, η οποία ανέλησε το κόστος και το κέρδος σε κάθε χώρα μέλος. Μπορώ αν θέλετε να το συζητήσω μαζί σας διμερώς και να σας δείξω και τα αποτελέσματα. Πάντως τα αποτελέσματα έλεγαν ότι η πρόταση αυτή είναι τέτοια ώστε να υποφεληθούν συνολικά όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες. Αυτό. Από εκεί και πέρα εσείς ε, θα αποφασίσετε αν ε, θέλετε να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση ή όπως είπατε πριν να κάνουμε κάτι άλλο. Σύντομα. Έχετε δίκιο πράγματι για αυτό το οποίο είπατε για το χρονοδιάγραμμα, αλλά αν δείτε το συμπέρασμα είναι πως ε, άρα δεν είναι απαραίτητο για αυτούς τους λόγους να εναρμονίσουμε σε επίπεδο ένωσης. Τέλος, σημείωσα αυτό το οποίο είπατε, πως ε, ε, Πράγματι ορισμένα δάνεια δίνονται μαζί με ασφάλιση, αλλά λέτε πως θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να επιλέγει άλλη ασφάλιση ο καταναλωτής, αλλά μετά του υπολογίζουν και άλλο επιτόκιο. Πράγματι έχετε καταθέσει μια σχετική τροπολογία. Πράγματι επίση, ε, ο κ. Φόξη και η Κομισιόν ανέφεραν τα του Ε, Θα ήθελα τώρα να απευθυνθώ προ την Κομισιόν να πω το εξή. Η διαγραφή των ε, πράξεων εξουσιοδότηση δεν σημαίνει δυσπιστία προς την ε, Κομισιόν, την εμπιστεύομαι, αλλά θεωρώ πως ο νομοθέτης ο ίδιος, εδώ δηλαδή το Κοινοβούλιο, δεν θα πρέπει να βγαίνει εκτός, θα πρέπει να λαμβάνει μόνος του δύσκολες τέτοιες αποφάσεις. Δεν είναι λοιπόν δείγμα δυσπιστίας προς την Κομισιόν. Καμιά φορά ε, αισθάνομαι πιο κοντά στην Κομισιόν παρά στο Κοινοβούλιο. Αλλά σας είπα, εδώ πέρα θα πρέπει ο νομοθέτης ο ίδιος να ε, είναι εγγυητής της ε, διαφάνειας. Ευχαριστώ και θα ήθελα να παρακαλέσω την γραμματεία λόγω της ώρας δεν βλέπω τώρα. Δεν έχω μπροστά μου τις ε, συνεδριάσεις. Να ξέρω πότε θα μπορέσουμε να το συζητήσουμε το ζήτημα για να έχουμε μια συνεδρίαση με τους κοιόδης ηγητές για να καταλέξουμε και σε κάποιες προθεσμίες. faire lettre à Madame Excusez-nous, on a un petit problème technique. Είχαμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα. Ε, υπάρχει ένα πρόβλημα για τις 5 Δεκεμβρίου που λέμε για την ψηφοφορία. Είναι πολύ μικρό το περιθώριο μετά γιατί στις 19 ή 20 Δεκεμβρίου ψηφίζουν οι προθεσμοί είναι πολύ σύντομοι, οπότε μια που οι σκιώδεις ζήτησαν να υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο, ε, προτείνω να στείλουμε μια επιστολή στην κυρία Μπόλ, που είναι πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, για να δούμε μήπως μπορούν εκείνοι να αναβάλουν την ψηφοφορία για τον Ιανουάριο. Συμφωνείτε? Οπότε έτσι μπορούμε εμείς και εμείς να ψηφίσουμε λίγο αργότερα. Μα δεν είναι μόνο για μένα. Ε, όλοι οι συνάδελφοι, όλοι οι συνάδελφοι το ζήτησαν. Γιατί δεν καταλαβαίνω δηλαδή και με τις τόσες τροπολογίες πώς ε, μπήκε τόσο σύντομα η προθεσμία. Ξέρετε κύριε Λεκτέρ, όλοι διαπιστώνουμε όπως και εγώ ότι ε, μερικέ φορέ, ενώ κανονικά χρειάζεται χρόνο, προσπαθούμε να πάμε γρήγορα, ενώ σε άλλα θέματα που χρειάζονται κατεπηγόντω αποφάσει, εκεί καθυστερούμε. Λοιπόν, εδώ θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και ελπίζω να πάνε όλα καλά. Σύντομη παρατήρηση. Μα εγώ δεν έχω πρόβλημα να κάνω με ένα κατάλογο ψηφοφοριών σύμπλην και να ψηφίσουμε. Αλλά δεν είναι αυτό το νόημα, έτσι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 Αγαπητοί συνάδελφοι, με ιδιαίτερη χαρά υποδεχόμαστε εδώ τον Επίτροπό μας, τον, Επίτροπο, τον Επίτροπο Μισελ Μπαρνιέ, ο οποίος θα μας παρουσιάσει κάτι πολύ βασικό για μας και μετά θα συζητήσουμε. Θα μας παρουσιάσει το πρόγραμμά του και το χρονοδιάγραμμά του για το έτος 2012, σχετικά με όλα τα κείμενα τα οποία πρόκειται να βγουν και τα οποία είναι θεμελιώδη τόσο για την εσωτερική αγορά, όπως και για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Θα δώσω λοιπόν το λόγο για 20 λεπτά περίπου στον Επίτροπο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους σας. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ μαζί σας και που μου δίνετε την ευκαιρία να αναφερθώ στον πίνακα αυτό που έχετε στα χέρια σας και που είναι το δικό μας νομοθετικό πρόγραμμα. Και να ξέρετε έτσι τι ακριβώ σημαίνει και πολιτικά. Ξέρω ότι μιλάω εδώ σε πολιτικού άντρε και γυναίκε που έχω εδώ μπροστά μου και ότι εσεί θέλετε πολλά από τα κείμενα αυτά, μια που δουλεύετε πάνω σε αυτά, είτε σαν εισηγητέ, είτε ω κοιόδη, είτε ω συντονιστέ και θέλετε όλα αυτά να τα γράψετε λοιπόν ε, στα πλαίσια της πολιτικής στιγμής μέσα στην οποία βρισκόμαστε. Ε, δεν θέλω να επαναλάβω ότι βρισκόμαστε μέσα σε μια πολύ σοβαρή κρίση για να μην πω κρίσεις, γιατί έχουμε πολλές κρίσεις να αντιμετωπίσουμε αυτή τη στιγμή. Την οικονομική, το δημόσιο χρέος, κοινωνικές δυσκολίες πολύ σοβαρές και άλλες πιο γενικές κρίσεις, αλλά και την κρίση εμπιστοσύνης που προστίθεται σε όλες τις προηγούμενες, κρίση εμπιστοσύνης από τους Ευρωπαίους πολίτες. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν θα έλεγα ότι επήγει οι Ευρωπαίοι ηγέτες να κάνουν αυτά που έχουν πει ότι θα κάνουν, αυτά που είπαν ότι ήθελαν να κάνουν. Για παράδειγμα, σκεφτόμαι εδώ τις αποφάσεις που λήφθησαν στις 26 Οκτωβρίου για να αντιμετωπιστεί η δημοσιονομική κρίση και η κρίση ε, δημόσιου χρέους. Και επίσης να κάνουν ε, και αυτά που πρέπει υπέρ της ανάπτυξης, διότι οι πολίτες περιμένουν να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να διευκολύνουμε την επιστροφή στην ανάπτυξη και στην απασχόληση. Και γι' αυτό ακριβώς θέλω, για άλλη μια φορά κυρία Πρόεδρε, να ευχαριστήσω τη δικιά σας Κοινοβουλευτική Επιτροπή που γνωρίζω καλά και πολλούς από εσά προσωπικά που βοηθήσατε γιατί βοηθήσατε πάρα πολύ όσον αφορά τις επιδόσεις της ενιαίας ε, πράξης. Ξέρουμε ότι είναι μια διαπίστωση μετά από την έκθεση του Λουί Κρές και την έκθεση στη συνέχεια του Μάριο Μόντι. Γνωρίζουμε ότι η μεγάλη ευρωπαϊκή αγορά, ο χώρος δηλαδή μέσα στον οποίο ζούμε όλοι μαζί, οικονομικός και κοινωνικός, αν λειτουργήσει καλύτερα, τότε όλες οι στρατηγικές ιδιωτικές, των επιχειρήσεων, των καταναλωτών, οι δημόσιες, της τοπικής αυτοδιοίκησης ή των περιφερειών ή των χωρών ή της ίδιας της Ευρώπης. Οι στρατηγικές αυτές λοιπόν, εφόσον η βάση, τα θεμέλια είναι στέρεα, τότε κάθε τέτοια στρατηγική θα πετύχει. Αυτό λοιπόν θέλουμε να πετύχουμε με αυτήν ε, την ε, νέα νέα πράξη. Υπάρχουν 12 κατά προτεραιότητα προτάσεις θέλουμε να πετύχουμε σε όλες και να έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις μέχρι τα τέλη της χρονιάς, εκτός από μία η οποία χρειάζεται περισσότερο χρόνο από νομική άποψη και που η συνάδελφός μου Νέλη Κρούς πρέπει να παρουσιάσει και έχει να κάνει με την ηλεκτρονική υπογραφή. Γι' αυτό το θέμα χρειαζόμαστε λίγο περισσότερο χρόνο. Πριν απαντήσω όμως στις ερωτήσεις σας και ακούσω πρώτα απ' όλα τι ερωτήσεις έχετε να μου κάνετε, θέλω να τονίσω λιγάκι τρεις προτεραιότητές μας. Όσον αφορά την ε, πράξη ενίας αγοράς, να ξέρετε ότι έχουμε κάνει τις δύο 12 αυτές προτάσεις, όπως μας ζήτησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δηλαδή τις ετοιμάσαμε για να εξεταστούν και να εγκριθούν όσο γίνεται πιο γρήγορα από το Συμβούλιο Υπουργών και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εξάλλου, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ζητήσω να ξανάρθω μετά από μερικές εβδομάδες εδώ, στην Επιτροπή σας, τις αρχές της επόμενης χρονιάς δηλαδή, για να ξεκινήσουμε με το δεύτερο στάδιο της πράξης για την ενιαία αγορά. Με το ίδιο πνεύμα δηλαδή, πολύ γρήγορα να περάσουμε στο δεύτερο στάδιο. Εγώ συνεργάζομαι με τους συναδέλφους μου και με τους άλλους επιτρόπους για αυτό το δεύτερο κύμα, το δεύτερο στάδιο της πράξης ενίας αγοράς. Γι' αυτό και θέλω να έχω τις δικές σας απόψεις και τις δικές σας προτάσεις. Σήμερα, εισαγωγικά, θέλω να επικεντρωθώ, όπως σας είπα, σε τρία ζητήματα. Πρώτον, η οικονομία υπηρεσιών, το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι δημόσιες αγορές. Πρώτα απ' όλα, οι υπηρεσίες οικονομίας. Πρώτα απ' όλα, εμείς θέλουμε να έχουμε μια καλή πολιτική για τις υπηρεσίες. Και είμαι λίγο επιφρακτικός μερικές φορές σε διάφορες ιδεολογικού τύπου δηλώσεις που λένε πριν αρχίσει να εφαρμόζεται η οδηγία για τις υπηρεσίες, πριν να την ξανανοίξουμε, πρέπει να μιλήσουμε για απορρίθμιση κλπ. Δεν έχω ξεχάσει τη συζήτηση που κάναμε την πρώτη φορά για την οδηγία για τις υπηρεσίες και θυμάμαι πάρα πολύ καλά όλες σας τις παρατηρήσεις. Δεν τα ξεχνά αυτά. Αυτό λοιπόν που τώρα εσείς πρέπει να ειστήσετε από τον Επιτροπό σας, από μένα δηλαδή, είναι η οδηγία αυτή να εφαρμοστεί καταρχήν καλά σε όλες τις, τις διαστάσεις. Αλλά ακόμα δεν είμαστε εκεί. Συνεπώς, προς το παρόν θα προσπαθήσω να εφαρμοστεί καλά η οδηγία αυτή, να υπάρχει η λεγόμενη ενιαία θηρίδα σε όλες τις ε, χώρες και στις περιφέρειες πολλές χώρες και όλα τα μέσα που προσφέρει η οδηγία αυτή να τεθούν σε εφαρμογή. Το ίδιο ισχύει και για την τρίτη οδηγία για τα ταχυδρομεία. Και εδώ θέλω να ενσωματωθεί ορθά στην εθνική νομοθεσία των χωρών. Λαμβάνοντας υπόψη τους χρήστες, έτσι, γιατί αποφάσισε να δημιουργήσω μία ομάδα χρηστών για την οδηγία την ταχυδρομική, έτσι ώστε να βεβαιωθώ ότι τίθεται σωστά και σε εφαρμογή. Η πρώτη ομάδα, η πρώτη συνάντηση μάλλον της ομάδας αυτής θα γίνει σύντομα για τα ταχυδρομεία. Έπειτα υπάρχει και η αμοιβαία αξιολόγηση της οδηγίας αυτής για τις υπηρεσίες. Να δούμε δηλαδή ποιες είναι οι επιδόσεις και να βεβαιωθούμε ότι όταν εφαρμόζεται η οδηγία αυτή δεν ε, βάζει τρικλοποδιά σε άλλου είδους ευρωπαϊκά κείμενα, σε άλλου είδους ενδεχομένω οδηγίες ή οτιδήποτε άλλο. Έχουμε μια φιλόδοξη στρατηγική πάντως για την αμοιβαία αυτή αξιολόγηση της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Ε, προσωπικά συναντήθηκα και με δημοσίους υπαλλήλους από διάφορες χώρες, εδώ και 1,5 χρόνο κάνω τον κύριο στις διάφορες χώρες. Πρόκειται να πάω σύντομα και στην Μάλτα και την Λετωνία και εκεί θα κλείσει ο κύκλος των επισκέψεών μου αυτών για να συζητήσω με τους δημοσίους υπαλλήλους το θέμα αυτό της αμοιβαία αξιολόγησης. Και κάτι ακόμα, τα επαγγελματικά προσόντα. Αυτό είναι το τρίτο σκέλος σχετικά με την οδηγία για τις υπηρεσίες. Το κείμενο το οποίο θα εξυγχρονιστεί πρέπει να συνεισφέρει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και να οδηγήσει σε μεγαλύτερη κινητικότητα σε πολλά επαγγέλματα. Σε αυτό το πνεύμα δουλεύουμε. Θέλουμε να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε όλες τις πτυχές της οδηγίας για τις υπηρεσίες, την αμοιβή αναγνώριση κλπ. Και όλα αυτά τα κάνω εξετάζοντας από πολύ κοντά μαζί με τα κράτη-μέλη τις ρυθμίσεις που ενδεχομένω να μην είναι κατάλληλες για το ένα ή το άλλο επάγγελμα. Και υπάρχει και ένα τέταρτο σκέλος που αφορά την οδηγία αυτή και που επέβαλα πρόσφατα στον κύριο Παρόσο για να ξεκινήσει η συζήτηση μεταξύ μας, αλλά ξέρω ότι και εσάς σας ενδιαφέρει, και αυτό είναι η σχέση που υπάρχει με τη βιομηχανία. Ο πρόεδρος Μπαρόσο έκανε μια παρουσίαση για την ανάπτυξη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Προάλλης και εκεί έδειξε ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα στην βιομηχανική βάση, όπου αυτή υπάρχει, και την οικονομία των υπηρεσιών που συνδέεται με τη βιομηχανία. Μιλάμε δηλαδή για θέσεις απασχόλησης που συνδέονται με την βιομηχανία αλλά που είναι στις υπηρεσίες. Και εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει πραγματικά δυνατότητα να επιστρέψουμε στην ανάπτυξη αν δεν έχουμε μια κατασκευαστική βιομηχανία η οποία θα προστατεύσει θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη. Δεν μπορεί η Ευρώπη μόνο να εισάγει ή να διαχειρίζεται προϊόντα τα οποία παράγουν άλλοι. Όχι, χρειαζόμαστε μια πραγματική βιομηχανική πολιτική. Ο συνάδελφος εξάλλου Ταγιάννη εντόπισε κάποιες τεχνολογίες κλειδί, τεχνολογίες του μέλλοντος, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας. Αν δεν αναλάβουμε εμεί την πρωτοβουλία για έρευνα στον τομέα αυτό, και αν δεν έχουμε επενδύσει στους τομείς αυτούς, τότε θα καταλήξουμε απλοί καταναλωτές κινέζικων και αμερικανικών προϊόντων. Όταν μιλάμε λοιπόν για την οικονομία των υπηρεσιών, να ξέρουμε ότι υπάρχουν υπηρεσίες άρρητα συνδεδεμένες με τη βιομηχανία. Η ύπαρξη ή μη των υπηρεσιών αυτών εξαρτάται από τη βιομηχανία. Θέλω βάσει της έκθεσης της κυρίας Κοράτσα Μπίλτ να περάσω στο θέμα των αθέμητων εμπορικών πρακτικών. Να ξέρετε ότι έχουμε συλλέξει πολλές πληροφορίες για τα συστήματα που εφαρμόζονται στα κράτη-μέλη προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο αθέμητος αυτός εμπορικός ανταγωνισμός. Και θα συνεχίσουμε την ανάλυση αυτή που κάνουμε με τα κράτη-μέλη και θα προτείνουμε, ελπίζω, μέσα στο 2012 συγκεκριμένα μέτρα. Και ένα τελευταίο θέμα στο οποίο θα αναφερθώ είναι η επικοινωνία. Τα παιχνίδια online. Συμφωνώ με την έκθεση Κρόιτσμαν για αυτό το θέμα και δουλεύω σε επίπεδο δράσης για να προχωρήσω στην προστασία των ανηλίκων. Με ενδιαφέρει επίσης το θέμα των αυθεντικών αγώνων, να μην υπάρχουν εκεί παρατυπίες. Και δεν αποκλείω βέβαια να πάω και ακόμα πιο μακριά μετά από αυτήν την πρώτη δράση που θα υποβάλουμε τον Ιούνιο και να προτείνουμε ρυθμιστικά μέτρα. Ελπίζω και το λέω εδώ ξεκάθαρα ε, μπροστά σας ότι θα προχωρήσω αναστάδια. Πρέπει να πάρουμε την πρωτοβουλία και πρέπει αυτό να το θέλουν όλοι και θα το προτείνω και στο Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έρχομαι στο δεύτερο κεφάλαιο στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ. Αυτό είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο. Θα είμαι σύντομο σε αυτό. Ξέρω πόσο πολύ σα ενδιαφέρει αυτό το σκέλο των υπηρεσιών που είναι υπηρεσίε και προ τον καταναλωτή που βελτιώνει και το διασυνοριακό εμπόριο. Ξέρουμε ότι το 2010-2011 Είχαμε το πολύ 9% των Ευρωπαίων πολιτών που έκαναν ε, διασυνοριακά αλλαγές, αγόρασαν δηλαδή αλλού από εκεί που μένουν. Είναι τεράστιες οι δυνατότητες που προσφέρει η αγορά αυτή. Θα κάνω λοιπόν ανακοίνωση από αυτού, εμπνεόμενος από τις εργασίες της ομάδας την οποία προεδρεύει ο κύριος ε, Αρία και να ξέρετε ότι και με την κυρία Κρούς και με άλλους συναδέλφους στην Επιτροπή προωθούμε τη δράση αυτή και τη δουλειά που γίνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις υπηρεσίες online. Το ηλεκτρονικό εμπόριο, ο εξυγχρονισμός της οδηγίας θα καλύψει πάνω σε αυτό ένα μεγάλο τμήμα. Οι υπηρεσίες online, τα κοινωνικά δίκτυα, τα διοικητικά θέματα online επίσης είναι μια εγκάρσια αντιμετώπιση που θα μας βοηθήσει σε διάφορους τομείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι συγκεκριμένοι, αλλά που αποτελούν μέχρι τώρα εμπόδιο στο online εμπόριο που έχει να κάνει με την πληρωμή, με την παράδοση, με την ενημέρωση των καταναλωτών, την κάλυψή του στην νομική και την διασυνοριακή προσφορά. Όλα αυτά τα θέματα θα τα δούμε στα πλαίσια της ανακοίνωσής μας αυτής για το online εμπόριο. Και τελευταίο σημείο, για να μην μακρύγορο είναι οι δημόσιες προμήθειες και δημόσιες αγορές. Ξέρω τις εργασίες της Επιτροπής σας. Ο Πρόεδρος σας ενδιαφέρεται όλος ιδιαίτερος και ο κύριος Ταραμπέλα, από ό,τι κατάλαβα, είναι υπεύθυνο για αυτό το θέμα. Θα είναι ένα συνολικό πακέτο μέσα Δεκεμβρίου, πριν τα τέλη της χρονιάς τέλος πάντων θα στο υποβάλω. Βέβαια με κάποια επιφύλαξη το λέω γιατί εξαρτάται από το πότε θα εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πάντως πρόκειται για τον εξυγχρονισμό και την απλοποίηση των κανόνων που ισχύουν για τις δημόσιες αγορές. Όπως επίσης για τις ε, ε, παραχωρήσεις και στα πλαίσια της Διεθνούς Συμφωνίας GPA που έχει να κάνει με τις δημόσιες αγορές, κάτι στο οποίο έχω δουλέψει με τον συνάδελφο Κάρλ Τεγκούχτ. Να πω και δύο λόγια για αυτές καθευτές τις δημόσιες αγορές. Η πρώτη μας ανησυχία είναι η απλοποίηση των διαδικασιών, γενικεύοντας την ε, διαδικασία να υπάρχει ε, των προτέρων διαπραγμάτευση, ποια είναι η τεκμηρίωση που απαιτείται, Πολλοί από εσά συμμετείχαν στη σχετική διάσκεψη και θυμόσαστε τι υπόθηκε εκεί, ότι είναι απαράδεκτο μερικέ μικρέ και μεσαίε επιχειρήσει να πρέπει να χρησιμοποιούν το 1 τρίτο του ποσού που ελπίζουν. Διακόπτε το μικρόφωνο του μιλτή. Ακούγεται τώρα πάλι. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε, να απλοποιήσουμε την τεκμηρίωση αυτή και να ξέρουμε ότι τελικά μόνο αυτός ο οποίος θα επιληχθεί θα πρέπει να παραδώσει όντως όλα τα έγγραφα έτσι όπως πρέπει. Περνάμε επίσης και στην ψηφιακή μορφή, η ηλεκτρονική υποχρεωτικά μερικές φορές, αντί να χρησιμοποιείτε χαρτί. Ή όπως κάνουμε και με το κούριελ. Ε, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, μειώνουν το διοικητικό άχθος. Και αυτό βοηθάει και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και αυτούς που έχουν να επιλέξουν. Θέλουμε να απλοποιούμε τη ζωή λοιπόν, χωρίς όμως βέβαια να μειώνουμε ε, την διαφάνεια καθ' άλλο, ούτε τον σωστό έλεγχο και τις σωστές διαδικασίες. Εδώ την ε, πρώτη φορά που ήρθα να μιλήσω για αυτά, σας μίλησα για τη φιλοδοξία μου και σας είπα ότι η αγορά αυτή γίνεται για όλους τους ανθρώπους, δεν γίνεται μόνο για, τους, τις μεγάλες επιχειρήσεις. Θέλουμε να αποφύγουμε όμως κάποιες απαιτήσει υπερβολικές οι οποίες δυσκολεύουν ε, τις μικρές και μεσές επιχειρήσεις και να οριοθετούμε βάσει ενός ε, ποσού τζίρου που θα αποτελεί την ε, απόδειξη για το σε τι βαθμό μπορεί να προχωρήσει σε μια συγκεκριμένη σύμβαση. Θέλουμε επίσης να διευκολύνουμε την πρόσβαση στους στις προσφορές και να φροντίσουμε τέτοιες προσφορές να μπορούν να κάνουν και οι πιο μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, να μην είναι μόνο οι μεγάλες. Όλα αυτά θα είναι ε, στην καρδιά της ανακοίνωσής μου, που θα περιλαμβάνει επίσης και τη διάσταση του περιβάλλοντος και την κοινωνική διάσταση. Σίγουρα οι αρχές που προτείνουν τους διαγωνισμούς πρέπει πάντα να είναι σε θέση να καλύπτονται. Αυτό όμως που προσπαθούμε να βρούμε είναι μέτρα τα οποία να βοηθούν στην αξιολόγηση του live ε, cycle cost που είναι ο πλήρης κύκλος ζωής ενός προϊόντος προς αγορά και να λαμβάνουμε υπόψη μας και τη διαδικασία παραγωγής του προϊόντος. Στην Παρασκευή οργανώσαμε μια διάσκεψη για την κοινωνική εταιρική σχέση από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ. Ήταν και πολλοί ευρωβουλευτέ στη διάσκεψη αυτή. Είχε μεγάλη επιτυχία. Για τις κοινωνικές επιχειρήσεις σίγουρα η απλοποίηση ε, όσον αφορά τις δημόσιες ε, προμήθειες είναι κάτι πολύ βασικό. Θα υποστηρίξουμε και την καινοτομία επίσης μέσω αυτής της νέας διαδικασίας για τις δημόσιες αγορές. Τέλος να πω κάτι για τις παραχωρήσεις που είναι κάτι πολύ βασικό όσον αφορά την εσωτερική αγορά της συμβάσεις παραχώρησης. Θέλουμε να συνεισφέρουμε, να προσφέρουμε νέες οικονομικές δυνατότητες στους Ευρωπαίους επιχειρηματίες. Ήδη η βάση παραχώρησης είναι κάτι πολύ σημαντικό σε διάφορες χώρες. 50% των υπηρεσιών στο τομέα των αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δίνονται βάσει της διαδικασίας αυτής συμβάσεων παραχώρησης στη Γαλλία ας πούμε. Πάνω από 10.000, πάνω από 80 δισεκατομμύρια ευρώ είναι με την διαδικασία αυτή. Δεν θέλω βέβαια, αγαπητοί ευρωβουλευτέ, να χρησιμοποιήσω άλλο, να προτείνω μάλλον άλλο ένα εργαλείο μέσα σε πολλά άλλα που διαθέτουμε. Όμως πιστεύω ότι είναι σημαντικά γιατί επιτρέπουν να έχουμε ένα ελαφρύ πλαίσιο, να είναι χρήσιμο, να υπάρχει εύκολος έλεγχος, να υπάρχει και ελαστικότητα στις τοπικές αρχές αλλά και έτσι διευκολύνονται ακόμα περισσότερο μικρομεσαίε επιχειρήσει για να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτέ τι συμβάσει παραχώρηση. Δεν θέλω νέου κανόνε, αλλά θέλω να διευκρινίσουμε πιο συγκεκριμένα τι ρυθμίσει που απορρέουν ήδη από τη συνθήκη. Θέλω δηλαδή να υπάρχει μεγαλύτερη νομική ασφάλεια και νομική βεβαιότητα. Μόνο έτσι αποφεύγουμε του κινδύνου διαφθορά ή κατάχρηση. Θα βελτιώσουμε έτσι λοιπόν την αποτελεσματικότητα των χρημάτων μας. Θα τα προστατεύσουμε. Κάτι ακόμα το οποίο απαιτεί δουλειά μέσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομικά και για τις εκθέσεις αντικτύπου είναι οι διεθνείς συμβάσεις. Πολλοί από εσά μου μίλησαν γι' αυτό, ότι μερικές φορές υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός, άδικος, όταν έχουμε διεθνείς συμφωνίες με δημόσιες συμβάσεις. Ορισμένε χώρες βλέπουμε ότι κλείνουν τις αγορές τους στις δικές μας επιχειρήσεις. Η Αμερική, για παράδειγμα, πρόσφατα το διαπιστώσαμε ότι προστατεύουν τις δικές τους επιχειρήσεις. Για μένα, η λύση δεν είναι να κλείσουμε το δικό μας χώρο, όχι, αλλά να βρούμε τα μέσα έτσι ώστε να υποχρεώσουμε ή να ενθαρρύνουμε τους άλλους με τους οποίους έχουμε σχέσεις να ανοίξουν τις αγορές τους. Παράλληλα, με εμά. Δεν πρόκειται για προστατευτισμό. Αυτό το κάνουμε και θέλουμε να το κάνουμε ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι άλλοι δεν ε, θα, παίρνουν, δεν θα προστατευτικά μέτρα για αυτούς, δεν θα προστατεύουν τις δικές τους τις αγορές. Γι' αυτό και θέλω να προτείνω ένα σχέδιο κανονισμού έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαθέτει ένα μέσο που να προσφέρει νομική βεβαιότητα και ασφάλεια και να φαίνεται έτσι στο δίκαιό μας ποιες είναι οι υποχρεώσεις μας και τι περιμένουμε σε διεθνέ επίπεδο. Αυτά. Την δυναμική αυτή θα την συνεχίσουμε με την πράξη ενίας αγοράς. Βλέπετε ότι υπήρχε μια αποκέντρωση των κειμένων, τώρα πιστεύω ότι οδηγούμεθα σε μια μεγαλύτερη συνοχή και έτσι θα μπορέσει να δουλέψει καλύτερα η βάση για την ε, οικονομία μας που είναι η μεγάλη και πραγματική ενιαία αγορά. Εξού και αυτή η πράξη που πιστεύουμε ότι θα μας θυμίσει ποια είναι τα θεμέλια μιας ε, ανταγωνιστικής ε, κοινωνικής οικονομίας που πολλές φορές ξεχνάμε. Το 2012 θα ξαναθυμηθούμε τα 20 γενέθλια της ενιαίας αγοράς. Δεν θα ήθελα να είμαστε μελαγχολικοί ούτε νοσταλγικοί επειδή βρισκόμαστε σε κρίση. Όχι, πρέπει να είμαστε γεμάτοι δυναμισμό γιατί η πράξη αυτή είναι μια ευκαιρία για να σκεφτούμε τα 21 αυτά γενέθλια, να δούμε τι πετύχαμε μέχρι τώρα με την εσωτερική ενιαία αγορά, αλλά να εντοπίσουμε και τα προβλήματα, ε, τις δυσκολίες, τις αδυναμίες και όπως κάναμε και στην Κρακοβία μαζί, να προσπαθήσουμε να δείξουμε με πρόσωπο ποιοι ε, νιώσαν επιτυχία από όλη αυτή τη διαδικασία. Αντίθετα, ποιοι δυσκολεύτηκαν, πού εντοπίζονται οι αδυναμίες. Μην ξεχνάμε λοιπόν τις δυνατότητες, τις ευκαιρίες που προσφέρει η ενιαία αγορά. Ε, θέλουμε να οργανώσουμε τον Οκτώβριο του 2012 μάλλον, επί τευκαιρίας 21ης αυτής επαιτίου της ενέας αγοράς, να οργανώσουμε έλεγα μία εβδομάδα όπου θα επικεντρωθούμε ακριβώς σε αυτά τα δυνατά και τα δύναμα σημεία της ενέας αγοράς. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. <laughs> Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε για το τόσο ε, σπουδαίο πρόγραμμα που μας παρουσιάσατε. Σίγουρα η επόμενη χρονιά θα είναι πολύ σημαντική. Τώρα, όπως είπατε και εσείς, λέω κι εγώ, να μην είμαστε νοσταλχικοί και θλιμμένοι τον ε, Οκτώβριο του 2012, και δεν θα είμαστε αν φροντίσουμε εμείς γι' αυτό και φροντίσουμε και πάλι για ανάπτυξη. Θα δώσω το λόγο στον πρόεδρο, τον κύριο Χάρμπορ, ο οποίος ήρθε για λίγο, έχει κάποιες ερωτήσεις, σίγουρα πολύ ενδιαφέρουσες, αλλά μετά θα πρέπει να μας εγκαταλείψει και πάλι. Ευχαριστώ, Μπερναντέτ. Ζητώ συγγνώμη από τον κύριο Επίτροπο που δίνει μου εδώ να τον καλωσορίσω. Και το τελευταίο σημείο το οποίο ανέφερε είναι ο λόγος για τον οποίο καθυστέρησα, γιατί εκπροσωπώ την Επιτροπή μας στον διάλογο τον νομοθετικό, τον διατλαντικό, καθώς θα έχουμε βεβαίω τη συνεδρίαση του Διατλαντικού Συμβουλίου την ερχόμενη εβδομάδα και βεβαίω υπάρχει, υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να απασχολήσουν το Συμβουλίο μας. Κάποια σχόλια τώρα θα έλεγα εξ ονόματος ολόκληρης επιτροπής. Πρώτα απ' όλα βεβαίως το πρόγραμμα σας ε, είναι καλοδεχούμενο. Υπάρχουν λίγες εκπλήξεις, λίγα πράγματα που δεν περιμέναμε, γιατί βεβαίως συνεργαζόμαστε ήδη στενά. Υπάρχουν πάρα πολλά χριστουγεννιάτικα δώρα τα οποία θα ξετυλίξουμε τα Χριστούγεννα και θα διαβάζουμε πάρα πολλούς μεγάλους φακέλους, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Θεωρώ όμως πως όσον αφορά τη μελλοντική μας συνεισφορά, η πρότασή σας να αρχίσουμε να αναπτύσσουμε ιδέες για τον δεύτερο γύρο της ε, νομοθεσίας της ε, κοινή αγοράς είναι πάρα πολύ θετικό και θα πρέπει να αρχίσουμε να προγραμματίζουμε ήδη. Το άλλο το οποίο θα ήθελα να επισημάνω, γιατί συμφωνώ μαζί σας πλήρως ότι πρέπει να δώσουμε ένα ανθρώπινο πρόσωπο στην ενιαία αγορά, όπως είπα στην Ολομέλεια και την προηγούμενη εβδομάδα. Η αγορά δεν είναι ένα, κάτι άψυχη κανόνες, είναι κάτι το οποίο βασίζεται στις επιτυχίες και τα επιτυχήματα ανθρώπων. Και βεβαίως ε, απαντήσατε στις ανησυχίες των πολιτών, κάτι για το οποίο γράφουμε τώρα μία έκθεση και ενδιαφέρον θα είναι να δούμε εάν μπορούν και άλλοι να... εάν μπορούμε να έχουμε κάποιες ενδιαφέρουσες απαντήσει σε αυτές τις ε, ανησυχίες και θα σας τα στείλουμε και εσάς για να υπάρξει κάποια συνέχεια. Βεβαίως δεν θα είναι νέα πολλά από αυτά τα πράγματα. Οπότε ο συντονισμός νομίζω των δραστηριοτήτων είναι κάτι το οποίο θα θέλαμε και εμείς προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε και άλλες επιτροπές ε, να δείξουν λίγη φαντασία και να ευλακούν μαζί μας την απάντηση αυτή. Ε, λυπούμε που δεν θα καθίσω να ακούσω τι απαντήσεις σας, ε, γι' αυτό και έκανα περισσότερο σχόλια, παλά ερωτήσεις. Τώρα λοιπόν θα πάω να στηρίξω ε, την Επιτροπή μας στον ε, υπερτλαντικό στον διάλογο με διατλαντικό των νομοθετών. Να ακούσουμε μια πρώτη σειρά ερωτήσεων καταρχήν και μετά θα απαντήσει ο Επίτροπος. Ο κύριος Βάμπη, κυρία Γκέμπχαρντ, Κρόσμαν και Ρούρλε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητέ Μισελ. Πρώτα απ' όλα σε ευχαριστούμε για την παρουσίαση και την προηγούμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια τα συζητήσαμε Θεωρώ λοιπόν πως ε, θα θέλαμε να δούμε κάποιες από αυτές τις προτάσεις σε έναν κανονισμό για να έχουμε γρήγορη εφαρμογή. Σήμερα όμως θα ήθελα να ρωτήσω τι γίνεται με την διαμόρφωση των προτάσεων περί δημοσίων προμηθειών ήδη ε, μας έχετε μοιράσει ένα έγγραφο. Είναι αυτό το πρόγραμμα. Θα λάβουμε ταυτόχρονα και τις τρεις προτάσεις και ταυτόχρονα έχουμε βεβαίως και την οδηγία ηλεκτρονικού εμπορίου όπου βεβαίως αναμένουμε και εκεί πέρα την πρόταση αυτή και αναρωτιόμαστε πότε θα έρθουν αυτές τις προτάσεις και όπως είπα εμείς θα θέλαμε ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των προτάσεων να είναι υπομορφή κανονισμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε κύριε Γκέμπαρτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε τον Μισελ Μπαρνιέ για αυτά τα οποία μας είπε. Θεωρώ πως πρέπει να προσέξουμε ε, κάτι το οποίο αναφέρθηκε στι εκθέσει Λουί Γκρέκ και Μάριο Μόντι. Να έχουμε δηλαδή μια συνολική προσέγγιση η οποία δεν θα χάνεται στην καθημερινή μα εργασία. Και νομίζω πω πράγματι αυτή τη στιγμή αυτή η συνολική έννοια της εσωτερικής αγοράς πρέπει να διατηρηθεί. Στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να αναφέρω λοιπόν δύο ζητήματα τα οποία υπάρχουν στα προγράμματα αλλά όχι ακριβώς όπως θα ήθελα εγώ. Το ένα είναι το θέμα των συλλογικών προσφύγων. Ξέρετε πως είναι απολύτως απαραίτητο να προχωρήσει η εφαρμογή του θέματος αυτού σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό θα πρέπει να προχωρήσουμε και να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός και όχι μόνο προπαρασκευαστικά έγγραφα. Το δεύτερο είναι μια απογοήτευση που έχουμε ένα κείμενο το οποίο είναι ήδη επιτάπητος και αφορά το δικαίωμα πρόσβαση των πολιτών σε τραπεζικό λογαριασμό. Υπάρχουν εκατομμύρια πολίτες που δεν έχουν τραπεζικό λογαριασμό παρά το ότι θα ήθελαν και έχουν δυσκολίες ήταν το ζήτημα, το είχαμε πει, λέγαμε θα κάνουμε ένα νομοθετικό κείμενο, τελικά κατέληξε να γίνει μόνο μια, κατέληξε να γίνει μόνο μια σύσταση. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω τι θα κάνετε στο μέλλον. Και εμάς ε, στην Επιτροπή Δικαιωμάτων Καταναλωτών είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Merci. Madame Ah, κυρία Ρουλε, όχι ο κύριος Κρούσμαν. Κρόιτσμαν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θέλω να κάνω τρεις παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα στηρίζω πλήρως την προσέγγισή σας πως είναι σημαντικό να παραμείνει η Ευρώπη ένας τόπος βιομηχανικός. Διαπιστώνουμε συνεχώς πως οι υπηρεσίες λειτουργούν όταν είναι κοντά στη βιομηχανία. Γι' αυτό πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα α, της Ευρώπης στην παγκόσμια αγορά. Τονίζω αυτό στην παγκόσμια αγορά. Δεύτερη παρατήρηση ε, αναφερθήκατε ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσον αφορά και στους διαγωνισμούς. Το χαιρετίζουμε αυτό και ακριβώς γι' αυτό θα θέλαμε να πούμε πως δεν θα πρέπει να αυξηθούν τα κατόφλια, είναι ήδη αρκετά υψηλά και ξέρετε πως πάρα πολύ, δύσκο, πάρα πολύ λίγες διασυνοριακές προσφορές υπάρχουν και θα μειωθούν κι άλλο και αυτές. Ξέρω βεβαίω πω αυτό το κάνουν τα κράτη-μέλη, θέλουν να διατηρήσουν τα μονοπόλια του, αλλά νομίζω πω ε, τα τωρινά κατόφλια είναι ιδανικά. Και τρίτον, χαίρομαι για το ότι η Κομισιόν ε, έχει υποβάλει ένα σχέδιο δράσης για το ζήτημα αυτό του τζόγου στο διαδίκτυο. Ξέρετε βεβαίως πως ε, εμείς με συντριπτική πλειοψηφία στην Επιτροπή μας και στο Κοινοβούλιο ήμασταν υπέρ και χαίρομαι και είμαι για το ότι θα έχουμε μία πρόταση η οποία θα είναι υποφελής για όλους, αμοιβαία υποφελής και θα πρέπει να στηρίξουμε την Κομισιόν στις ε, προτάσεις της. Ευχαριστώ. Merci, Monsieur πρέπει να είμαι σύντομη γιατί και εγώ θα πρέπει και μισή να φύγω. Λοιπόν, χαιρετίζω το πρόγραμμά σας. Είπατε πως για τον εξυγχρονισμό τη αμοιβαίας αναγνώριση. θα πρέπει να δούμε τα ρυθμισμένα, τα κλειστά επαγγέλματα. Να πω πως ε, πράγματι υπάρχουν ε, αρκετοί φόβοι γιατί ειδικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις υπάρχει ο φόβος πως τα ρυθμισμένα αυτά επαγγέλματα θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κάποιες παρεξηγήσεις όσον αφορά την ε, διπλή εκπαίδευση και όσον αφορά το ζήτημα των, ε, της ε, των επαγγελματικών προσόντων. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια ισοτιμία. Μια δεύτερη παρατήρηση. Είδαμε χαρά πως ε, αναφέρατε το ζήτημα των ηλεκτρονικών δημοσίων προμηθειών, αλλά λυπούμε κάπως για το ότι διαχωρίστηκε από τις υπόλοιπες μεταρρυθμίσεις και λέτε πως θα έρθει το 2012. Εγώ θεωρώ πως αν έχουμε μια πραγματική μεταρρύθμιση των δημοσίων προμηθειών πρέπει να ληφθεί υπόψη και ε, η ηλεκτρονική προκήρυξη. Και θα πρέπει η εξ εξερχής να συμπεριληφθεί. Νομίζω πως είναι αναγκαίο αυτό. Ευχαριστώ. Madame Monsieur le Σα ευχαριστώ. Ο κύριος Επίτροπος θα απαντήσει τώρα σε αυτή την πρώτη σειρά ερωτήσεων και έπειτα υπάρχουν πολλοί που έχουν ζητήσει το λόγο. Θα σας δώσω το λόγο λοιπόν στον καθένα για ένα λεπτό έτσι ώστε να μπορέσει να απαντήσει ο επίτροπο σε όλους. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κατάλαβα καλά τη λόγω αποχώρηση του Μάλκομ Χάρμπορ και θα ήθελα ίσως να διευκρινίσω ότι κατά τη γνώμη μου, και το έχω πει επαναλημμένως, αλλά νομίζω και εσείς το ίδιο πιστεύετε, το, η πράξη νέα αγορά έχει δύο χαρακτηριστικά. Καταρχήν είναι συλλογική για 10 επιτρόπους, όχι μόνο για ένα κείμενο, αλλά και για ένα πρόγραμμα για την ανάκαμψη ολόκληρης της ενίας αγοράς. Για σας, ως Επιτροπή ΜΚΟ, βέβαια είστε αρμόδια για αυτήν την υπόθεση, αλλά υπάρχουν και άλλες επιτροπές που συλλογικά ασχολούνται με το θέμα, όπως και εγώ με τους 10 συναδέλφους, και είναι σημαντικό εδώ να διατηρηθεί αυτή η συνοχή ανάμεσα σε όλες τις επιτροπές που εργάζονται για αυτήν και για, ανάμεσα στους επιτρόπους, αλλά και με το ε, Συμβούλιο των Υπουργών. Και έπειτα είναι μια διαρκής διαδικασία που συνεχίζεται και γι' αυτό μίλησα για δεύτερη φάση. Μπορεί να είναι νόμοι, οδηγίες, κανονισμοί, άλλες πρωτοβουλίες. Εγώ θα ήθελα από κοινού να σκεφτούμε αυτή τη δεύτερη φάση για να συνεχιστεί ως, όπως είπαμε, αυτή η διαδικασία της ενίας αγοράς. Έχουμε πολλά κείμενα που φτάνουν στα τέλη του χρόνου και αυτό είναι πολύ ικανοποιητικό αλλά και λίγο ε, ενοχλητικό γιατί ε, ε, μπερδεύονται όλα μεταξύ τους. Ε, και εσείς κύριε ε, δώσατε μια πιο προοδευτική εικόνα σε αυτό το πρόγραμμα. Να επιβεβαιώσω ότι το πακέτο δημόσιες προμήθειες καταρχήν σημαίνει την, την εξαρχής εξέταση αυτών των ε, δημόσιων αγορών. Δεύτερον, έχουμε τις συμβάσεις παραχώρησης ε, και θα έρθει το πακέτο αυτό γύρω στα μέσα Δεκεμβρίου. Ίσως να λείπει ακόμα, μια, να υπάρχει μάλλον ακόμα μια βεβαιότητα για την αγορά DPA, αλλά έχουμε αποφασίσει με τον κύριο Τεγκούχτ να προχωρήσουμε γρήγορα, αν όχι τον ίδια στιγμή με τα άλλα θέματα, αλλά αμέσως μετά. Επίσης, λόγω συμφόρησης για, στις υποθέσεις της Κομισιόν και για να είναι πιο ανάγνωστα τα θέματα και που συμφωνήσαμε με την ομάδα να διαφοροποιήσουμε λίγο την ανακοίνωση του e-commerce αρχές Ιανουαρίου παρά 20 Δεκεμβρίου με ένα πακέτο κειμένων που κανένας πια δεν θα καταλαβαίνει τίποτα και θα τα παρουσιάσουμε όλα μαζί. Εγώ ίδιος νομίζω πως σε ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως το e-commerce θα το συζητήσω με τους συναδέλφους για να δούμε μήπως μπορούμε αυτό να το κάνουμε αρχές Ιανουαρίου για να γίνει πιο κατανοητό. Συμφωνώ και με τον Ανδρέα Ζαρβάμπα για την ιδέα ότι όσο περισσότερο προχωρήσουμε με μηχανισμού, τόσο καλύτερα. Μάλλον αυτό όμω δεν είναι πάντα η άποψη του Συμβουλίου των Υπουργών, αλλά εν πάση περιπτώσει για το διεθνέ επίπεδο, για το GPA, κανονισμό θα προτείνουμε με τον κύριο Τιγκούχτο, όπω το κάνουμε γενικά κάθε φορά που μπορούμε να το κάνουμε στο άλλο τμήμα του χαρτοφυλακίου μου για τους ε, κανονισμούς, τους ε, χρηματοπιστωτικούς. Αυτά είχα να πω στον Αντρέα Σβάμπ. Η Εύελιν Γκέμπαρτ μίλησε για μια σφαιρική προσέγγιση. Θα πρέπει να αποφύγουμε ένα διπλό ε, κατακαιρματισμό. Κατακαιρματισμό ανάμεσα στις διάφορες προτάσεις για να μείνουν συνεκτικές και γι' αυτό θα ήθελα να πάρει ζωή η πράξη νέας αγοράς, ε, να επιβεβαιώνεται κάθε χρόνο πέρα από τις δημόσιες διεκδηλώσεις που μπορούμε να κάνουμε, να δείχνουμε δηλαδή ότι κάναμε αυτό που είπαμε και να υπάρξει ένα νέο κύμα προτάσεων σε αυτή τη νέα φάση. Και δεύτερη δε, ε, ο δεύτερος κατακαιρματισμός που πρέπει να αποφευθεί είναι εντός της Ένωσης ανάμεσα, και το λέω αυτό ειλικρινά, γιατί είναι άλλωστε και επίκαιρο το θέμα, ανάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης και για τις υπόλοιπες. Ορισμένες χώρες θέλουν να προχωρήσουν πιο πολύ να κάνουν ε, διακυβέρνηση. Άλλοι που δεν ήθελαν να μπουν στην Ευρωζώνη θα το μπορούν να το κάνουν όταν θέλουν. Πάντως η Ευρωπαϊκή, η, μάλλον η ενιαία αγορά αποτελείται από τους 27. Και αυτή είναι και η δύναμη της. Και το λέω εδώ, στο Παρίσι, στο Λονδίνο, στο Βερολίνο και στις άλλες πρωτεύουσες ότι υπάρχει μόνο μία ενιαία αγορά και εργάζομαι για κανονισμούς, νομοθεσίες και πρόοδο γενικότερα για το σύνολο της ενιαίας αγοράς, γιατί διαφορετικά είναι μια ενιαία αγορά των χρηματοπιστωτικών ε, ε, υπηρεσιών που δεν υπάρχει ακόμα και γι' αυτό και προσπαθώ να αποφύγω τον κατακαιρματισμό. Για τις συλλογικέ προσφυγές. Δύο πρωτοβουλίες υπάρχουν για τους καταναλωτές. Ο εναλλακτικός κανονισμός για τις... Μάλλον, εναλλακτικός διακανονισμός των διαφορών. Αυτό το κείμενο θα παρουσιαστεί τέλη του μήνα, τώρα του Νοέμβρη. Και όσον αφορά τις λογικές προσφυγές, όπως είπε και η κυρία Ρέντινγκ και ο κύριος Αλμούνια, εργάζονται από αυτόν ε, πολύ δραστήρια για τους επόμενους μήνες. Δεν μπορώ να πω ακριβώς ποια είναι η προθεσμία όπου θα είναι έτοιμο το κείμενο, αλλά θα το ζητήσω να σας απαντήσουν. Ξέρω τώρα ότι την ανησυχία σας για τους, για τους βασικούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Εγώ ο ίδιος ε, θέλησα να δώσω χρόνο για τις συμβάσεις. Είπα επίσης στις τράπεζες ότι αν δεν σημειωθεί πρόοδος μέσω των ε, βολονταριστικών πολιτικών των κρατών μελών, εμείς θα νομοθετήσουμε. Κυλά ο χρόνος λοιπόν και ξεκινάμε με μία τέτοια βασική, 30, ε, βασική ιδέα, 30 εκατομμύρια κόσμος δεν έχουν τραπεζικό λογαριασμό και μάλιστα τους αρνούνται την δυνατότητα να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό. Ε, έτσι λοιπόν, Νομίζουμε ότι πρέπει να υπάρξει πρόσβαση στους βασικούς ε, λογαριασμού, σε έναν βασικό λογαριασμό και αν τα κράτη-μέλη δεν κινηθούν, εμείς θα, θα προτείνουμε μέχρι πριν το τέλος του 12 ε, σε νομοθεσία. Και κάτι ακόμα συνδέεται με αυτό εδώ και δεν θέλω να αφήσω να περάσει προθεσμία, είναι το θέμα της διαφάνειας των τραπεζικών εξόδων. Υπάρχουν κόστη ανεξήγητα και μυστηριώδη που συχνά επιβάλλονται στους ε, πελάτες των τραπεζών, ιδιαίτερα με τη χρήση των τραπεζικών καρτών και ζήτησα διαφάνεια. Και εδώ με το πνεύμα της ε, συνεργασίας και όχι της επιβολής είμαι απογοητευμένος με την απάντηση που, δεν πήρα μάλλον από τις τράπεζες και μέσα στο 2012 θα προτείνουμε σχετική νομοθεσία. για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στα θέματα αυτά και μεταξύ των οποίων και του τραπεζικού λογαριασμού. Αλλά καταλαβαίνω την ανησυχία σας, αλλά σίγουρα θα περάσει καιρός, ε, θα προχωρήσουμε ε, εάν δεν έχουμε ε, σωστές και πιστικές αποφάσεις από πλευράς, προτάσεις μάλλον από πλευράς του τραπεζικού τομέα και των κρατών μελών. Τώρα, Είπατε ότι είναι σημαντικό να υπάρξει βιομηχανία, αλλά σημαντικό είναι να υπάρχει νέα βιομηχανία, μόνο που πολλές χώρες έχουν εγκαταλείψει τη βιομηχανία τους. Και οι χώρες ε, οι οποίες έχουν επιλέξει το πρότυπο του εμπορίου και των υπηρεσιών, των συναλλαγών, των εισαγωγών, αντί να έχουν ή να κατασκευάσουν βιομηχανική βάση, είναι αυτές που έχουν και τα μεγαλύτερα χρέη αυτή τη στιγμή. Είναι λογικό. Και εδώ λοιπόν θα πρέπει να αποκομίσουμε διδάγματα από την κρίση. Δεν υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, αποδοτική οικονομία χωρίς ισχυρή βιομηχανία. Βεβαίως όλα τα μέτρα του, της πράξης την νέα αγορά λαμβάνονται για να διευκολύνουν τον βιομηχανικό ιστό. για να επιβεβαιώσω ότι εργάζομαι δραστήρια στο πνεύμα της ε, συζήτηση που είχαμε πριν από κάποιες μέρες ε, στο Στρασβούργο για το πρόγραμμα δράσης για το online εμπόριο. Η κυρία Ρούλε μίλησε για τα κλειστά επαγγέλματα και είπα ότι δεν είναι μόνο το θέμα των κλειστών επαγγελμάτων, μάλλον ο αριθμός τους που δημιουργεί πρόβλημα, είναι η ανάλυση που πρέπει να κάνουμε αναχώρα. γιατί έχει απλοποιηθεί από εθνικά μέτρα ένας αριθμός επαγγελμάτων και υπάρχουν ένα σωρό φραγμοί επιδεσμεύσεις που δεν είναι δικαιολογημένοι και ακριβώς θα δουλέψουμε για κανθένα από αυτά τα επαγγέλματα και θα σας υποβάλουμε συγκεκριμένες, ε, θα υποβάλουμε μάλλον στα κράτη-μέλη συγκεκριμένες προτάσεις. Ε, τώρα, οι ηλεκτρονικές δημόσιες ε, προμήθειες και αυτό είναι κάτι για στο οποίο πιστεύω είναι τμήμα του γενικού πακέτου και αργότερα, αλλά όχι πολύ αργά, θα κάνουμε μια ανακοίνωση για να δώσουμε την συνέχεια και για να ανακοινώσουμε τις πρακτικές των κρατών μελών. Σα ευχαριστούμε κύριε Πίτροπε. Πολύ σύντομα, γιατί εγώ δεν θα ξαναπάρω το λόγο, γιατί είναι πολλοί αυτοί που θέλουν να πάρουν το λόγο. Θέλω να προσθέσω τα όσα είπατε για την πρόσβαση στι ε, τραπεζικέ υπηρεσίε. Σε αυτή τη φάση αβεβαιότητας και αφιβολίας των πολιτών για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, εδώ μπορούμε να καθησυχάσουμε κάποιου ε, συμπολίτε μα ιδιαίτερα του πιο εύθραυστου, και να του ενσωματώσουμε σε αυτή τη ζωή τη εσωτερική αγορά, να μην μείνουν στην άκρη δηλαδή, σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Θα δώσω το λόγο για ένα λεπτό τώρα στους υπόλοιπους που θέλουν να υποβάλουν ερωτήσεις. Βαντεκάπα. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Έχω δύο ερωτήματα. Το πρώτο, για να έχουμε και αν έχουμε πλήρη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς θα έχουμε μία αύξηση ε, του ΑΕΠ ε, τουλάχιστον κατά 10%. Ε, τι κάνετε πέρα από τη νέα νομοθεσία για την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας. Έχετε επαρκείς πόρους δεύτερον. Καμία πρόταση για την πνευματική ιδιοκτησία. Υπάρχουν διάφοροι φάκελοι εδώ πέρα σε εσά και στους άλλους επιτρόπους γιατί το 2012 δεν θα έχουμε νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία ε, από εσάς, αν κατάλαβα καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Επίτροπε. Εάν ε, μου επιτρέπετε θέλω να σας μιλήσω σου ειδικά για ένα θέμα το οποίο δεν αναφέρατε. Σημειώνω πως του χρόνου, το δεύτερο εξάμεινο, η Κομισιόν θα καταθέσει την Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τον καταναλωτή. Και θα ήθελα άρα να σας θέσω ορισμένα ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα στις κοινωνίες μας έχουμε πολύ περισσότερη διαφήμιση. Ε, διαφήμιση που στοχεύει επίσης και τα παιδιά στα ΜΜΕ, στο ίντερνετ κτλ. Αναρωτιόμουν αν η Κομισιόν θα συμπεριλάβει και αυτή την τυχή διαφήμιση που στοχεύει τα παιδιά. Δεύτερον, Διαφήμιση για τα υνοπνευματώδη προϊόντα. Μιλάμε για social media κτλ. Μην ξεχνάτε πως τα παιδιά ιδιαίτερα ασχολούνται με αυτά. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μια στρατηγική όσον αφορά ακριβώς τη διαφήμιση των υνοπνευματοδών στο διαδίκτυο. Θα Έχετε λοιπόν αυτή την πτυχή στο πρόγραμμά σας. Νομίζω πως οι οργανώσεις των καταναλωτών πρέπει να λάβουν μέρος σε αυτή τη διαδικασία. Ελπίζω να εξυπακούεται για την Κομισιόν και αυτό δεν το είπατε. Ευχαριστώ. Κύριε Ριγκογέν. Muchas gracias, comisario. Σας ευχαριστούμε, Επίτροπε. με τα αρχικά σας λόγια ότι πρέπει δηλαδή να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη, αλλά πρέπει κυρίως να δεσμευτούμε για να σεβαστούμε αυτά που είπαμε ότι θα κάνουμε. Κατά συνέπεια, σε αυτή την πρόταση για το πρόγραμμα εργασίας 2012 δεν υπάρχουν νομοθετικές προτάσεις σε σχέση με την ανάπτυξη ε, ταμείων αλληλέγγυων επενδύσεων. Γιατί υπάρχει αυτή η έλλειψη, ενώ μιλάμε για προτεραιότητα, για την πράξη νέα ε, αγορά, για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη και να υπάρξει ανάκαμψη. Μιλάμε για επίγον μέτρο δεδομένη τη ε, ισχύουσα οικονομική κατάσταση. Κύριε Πίτροπε, λοιπόν, πότε προβλέπετε να υποβάλλετε αυτό το ευρωπαϊκό πλαίσιο για το Ταμείο Αλληλέγγυων Επενδύσεων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θα κάνουμε άλλη μια σειρά ερωτήσεων σύντομα για να μπορέσει να μας απαντήσει ο Επίτροπος πριν να φύγει. Κυρία Κοράτζα Μπίλτ, ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Χαίρομαι και σας ευχαριστώ για την δέσμευσή σας που θα ήθελα που μάλιστα το συζητήσατε μαζί μας στο ΕΛΚ για την ε, ψηφιακή αγορά την ψηφιακή Ευρώπη αναφέρεται μια ολόκληρη σειρά δράσεων, ενεργειών, αλλά το ερώτημά μου είναι τι θα κάνετε για να αντιμετωπίσετε πραγματικά την, τους δισταγμούς, των επιφύλακ, της επιφύλαξης που υπάρχουν στο κράτη τον προστατευτισμό που υπάρχει, γιατί δεν θέλουν να δώσουν την ίδια αξιοπρέπεια, το ίδιο καθεστώς στη ε, μετακίνηση, στη κυκλοφορία αγαθών ε, ψηφιακά υπάρχουν προβλήματα με την πνευματική ιδιοκτησία κτλ. κτλ. Ε, είναι επίσης το σχέδιο δράσης για το εμπόριο, για το οποίο εργάζομαι αυτή τη στιγμή, που έχει προβλεφθεί για την αποτελεσματικότητα του εμπορίου και θέλω να δω για τη... πώς αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο της, της πράξης της νέα αγορά και θέλουμε να δούμε τους εταίρους να, που να δεσμεύονται και να αναλαμβάνουν πραγματικά τις ευθύνες τους. Γι' αυτό θα πρέπει να διατηρήσουμε αυτή την πορεία, αυτή την ορμή για να μπορέσουμε να κλείσουμε μέσα στον επόμενο χρόνο. Ευχαριστώ κύριος Μάγερ. Ευχαριστώ κύριε Πίτροπα. Ε, βεβαίως ε, μπορώ να στηρίξω αυτά τα οποία είπατε. Βεβαίως πράγματι έχουμε την εσωτερική αγορά, έχουμε τις ε, τέσσερις ελευθερίες, αλλά βεβαίως δεν λειτουργεί, γι' αυτό χρειαζόμαστε το χ και το ψ. Αλλά το συζητήσαμε και πριν έρθετε αυτό το οποίο δεν υπάρχει και δεν υπήρχε από την αρχή, ήταν η εφαρμογή αυτών των οποίων αποφασίζουμε στις χώρες. Δεν έχει νόημα να μιλάμε εμείς εδώ πέρα για συλλογικές προσφυγές, αναλλακτικέ ε, δυνατότητες ε, επίλυσης διαφόρων και να μην λειτουργεί τίποτα. Το δεύτερον, πρέπει να προσέξουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα τρία βασικά επίσης θεσμικά όργανα, να μην κάνουμε μόνο απλώς νόμους. Τα κράτη δεν πρέπει να ε, ασχολούνται μόνο με το Συμβούλιο, αλλά και στα εθνικά τους κοινοβούλιο. Και στη Γερμανία το ίδιο. Είχαμε τη συζήτηση επίσης για το Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Συμβάσεων, όπου υπάρχει άποψη πως είναι κάτι το καινούριο, το οποίο μας αφαιρεί δικαιώματα κτλ. Παρά το ότι ε, είναι πράγματα τα οποία κατ' ουσίαν έτσι είναι υφιστάμενο δίκαιο. Οπότε θεωρώ πως χρειάζεται περισσότερη ενημέρωση στα κράτη-μέλη και στα, στην ομοθετική εξουσία εκεί πέρα για το τι κάνουμε εδώ πέρα, για να μην θεωρούν πως συνεχώς τους παίρνουμε εθνική κυριαρχία. Γιατί αυτά τα οποία κάνουμε είναι ήδη πράγματα αποφασισμένα και εμείς απλά τα εφαρμόζουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Σας ζητώ πραγματικά να τηρείτε το χρόνο σας, γιατί ο Επίτροπος δεν θα έχει το χρόνο να απαντήσει διαφορετικά. Κύριος Αντώνιο Κορέια Ντεκάμπος. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Μια ερώτηση ενός λεπτού. Γιατί δεν θα έχουμε του χρόνου μια ανακοίνωση για τις υπηρεσίες γενικού ε, μάλλον κοινο, ε, γενικού συμφέροντος, μιλήσατε για ανακοίνωση για τις συμβάσεις παραχώρησης, δημόσιες και ιδιωτικές και ίσως και για τις δημόσιες-δημόσιες συμβάσεις παραχώρησης. Επί, μας, είχατε μας υποσχεθήκατε κάτι για τις κατοικές ενισχύσεις και πολύ καλό είναι αυτό γιατί είναι απαραίτητο να γίνει. Αλλά και μάλιστα μιλήσατε για το ηλεκτρονικό εμπόριο, για τις δημοσιοκρατικές προμήθειες, για τις ηλεκτρονικές προμήθειες, όλα αυτά πολύ ωραία και καλά. Ακόμα και για τα τυχερά παιχνίδια online. Δεν είμαι πορτανός, αλλά εν πάση περιπτώσει δέχομαι ότι πρέπει να ρυθμιστεί το ζήτημα. Αλλά για την ε, κοινωνική οικονομία ανταγωνιστικών αγορών, όταν μιλήσατε γι' αυτό, είμαι λίγο απογοητευμένος γιατί δεν βλέπουμε τίποτα για τις υπηρεσίες και γενικού οικονομικού συμφόρτου. Ευχαριστώ πολύ. Σύντομα, κυρία Βάις Γκέρμπερ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Επίτροπε. Κύριε Μπαρνιέ, στηρίζω διάφορες δικές σας προτάσεις στο δημοσιονομικό τομέα κυρίως, αλλά υπάρχει και μία με την οποία δεν συμφωνώ πολύ. Πρόκειται για τις συμβάσει παραχώρησης της υπηρεσίας. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται τέτοια οδηγία. Το Κοινοβούλιο έχει αποφανθεί και έχει πει ότι πρέπει πρώτα να φανεί ότι υπάρχει στρέβλωση της εσωτερικής αγοράς. Οπότε ρωτάω, υπάρχει? Υπάρχει έπειτα τέτοια τεράστια δυνατότητα διασυνοριακά, γιατί παίζει και το θέμα της εμπιστοσύνης σε θέματα που έχουν να κάνουν με το νερό, για παράδειγμα, με τα απόβλητα. Ρωτάω, υπάρχουν πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θέλουν να πάνε στο εξωτερικό. Πολλές συμβάσεις είναι μακροχρόνιες. Η κατασκευή μιας γέφυρας, για παράδειγμα, κρατάει 10-15 χρόνια. Άρα η σύμβαση είναι μακροχρόνια. Γι' αυτό και λέω ότι εδώ δεν χρειάζεται απαραίτητα μια ευρωπαϊκή οδηγία, γιατί μόνο γραφειοκρατία θα προσθέσει. Μπορείτε και αλλιώ να αντιμετωπίσετε την διαφθορά, όχι μόνο μέσα από μια τέτοια οδηγία. Πρόεδρος, Μπάρβαρα Βέιλερ τώρα. Ευχαριστώ. Δεν θέλω εγώ να μιλήσω για αυτό το σημείο, αλλά να επανέλθω λιγάκι σε αυτά που είπε ο Δ. Μάγερ. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να μην ξεσκώνουμε πολύ, να μην περιμένουμε πολλά ε, πράγματα. Για, ε, να τα λύσουν τα κράτη-μέλη. Γιατί κάνουν ματιρές οικονομίες τα κράτη-μέλη, μειώνεται η αγοραστική δύναμη των πολιτών, γι' αυτό θα πρέπει να μην έχουμε πάρα πολύ μεγάλες προσδοκίες. Είναι ευαίσθητο αυτό το θέμα. Δεύτερο, η εναλλακτική επίλυση διαφορών, ναι εντάξει τη θέμε, είναι σημαντική, αλλά δεν αντικαθιστά την συλλογική προσφυγή. Δύο πράγματα διαφορετικά συμπληρωματικά. Τελευταίο, πρωτοβουλία για τα τρίτα κράτη. Τι θα είναι αυτό, ανακοίνωση, ε, πρωτοβουλία, τι ακριβώς θα είναι, για πείτε μας λίγα παραπάνω γι' αυτό. Τελευταία, κύριε Σαλτεμόζερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και κύριε Επίτροπε. Υπάρχουν πολλές καλές πρωτοβουλίες και χαίρομαι που βλέπω ότι για τα παιχνίδια online Τελικά εισακούστηκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μας ακούσατε και αποφασίσετε να ενισχύσετε την συνεργασία μεταξύ των χωρών μελών πριν οδηγηθείτε σε νομοθεσία. Θέλω όμως να επανέλθω λίγο σε αυτό που είπε η Μπάρμπαρα Βάιλερ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη σκεφτεί με ποιο τρόπο εμείς στην εσωτερική αγορά θα διασφαλίσουμε μια βελτίωση των ε, ήδη υπαρχουσών ρυθμίσεων αυτό το aiming and shaming, εντάξει, από τη μια μεριά. Από την άλλη μεριά όμως, δεν έχουμε χρόνο τελικά με όλες αυτές τις ε, συνθήκες. Πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε τους κανόνες στην εσωτερική αγορά και έτσι θα έχουμε πιο θετικές συνέπειες και μια αγορά που θα λειτουργεί πολύ καλύτερα. Θέλω να το σκεφτούμε αυτό. Ευχαριστώ. Πολλές ερωτήσεις κύριε Επίτροπε πολλές ερωτήσεις και σίγουρα θα έχετε λίγο χρόνο για να απαντήσετε. Σας ακούμε. Θα προσπαθήσω να είμαι και συγκεκριμένος και σύντομος. Για τον κύριο Βαντερκάμπ. Υπάρχει ένα νούμερο το οποίο με εξέπληξε σχετικά με την ανάπτυξη που μπορούμε να βρούμε στην εσωτερική αγορά εφόσον αυτή λειτουργεί καλά. Οι αναλύσεις μας και ορισμένοι λένε ότι είναι υπερβολικά ε, αισιόδοξε θα είναι 2 με 4% παραπάνω αν λειτουργούσε καλύτερα, αν λειτουργούσε καλά η εσωτερική αγορά. Ήδη το 2-3-4% παραπάνω ανάπτυξη ε, ε τη σήμερα ημέρα καταλαβαίνετε πόσο χρήσιμο θα ήταν. Εμείς έχουμε μια διτή ανησυχία. Πρώτον, εφαρμόζεται καλά ότι οι διατάξεις έχουν ήδη ψηφιστεί και απ' την άλλη οι νέες αυτές ε, προτάσεις να προχωρήσουν. Επίτηδες κύριε Βαντερκάμπ δεν αναφέρθηκα στην ε, πνευματική ιδιοκτησία. Γιατί είναι κάτι που παρακολουθεί περισσότερο η Επιτροπή Τζούρι εδώ στο Κοινοβούλιο. Αλλά σας διαβεβαιώνω ότι θα υπάρχουν πολλές προτάσεις το 2012 όσον αφορά την πνευματική ιδιοκτησία. Για τα δικαιώματα ε, πνευματικής ιδιοκτησίας των δημιουργών και θα φροντίσουμε να διευκολύνονται οι συναλλαγές και εκτός συνόρων. Έπειτα υπάρχει και η πράσινη βίβλος για το οπτικοακουστικά. Το 2012 λοιπόν θα έρθουν πολλά πράγματα και τα πνευματικά δικαιώματα. Για την κυρία Ανχέντ, αναφερθήκατε σε πράγματα που εμένα με νοιάζουν πολύ και έχουν να κάνουν με την κοινωνία. Κύριε Κρότσμαν, και η Σαλτεμόζερ. Υπάρχουν θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την κοινωνία, με τους νέους, με τον εθισμό, με την ε, προστασία των ανηλίκων, ε, το θέμα των παιχνιδιών online, το θέμα των καταχρήσεων από τις διαφημίσεις ή το θέμα της κατανάλωσης αλκοόλ. Όλα αυτά είναι βέβαια στην αρμοδιότητά μου και αυτό που με ενδιαφέρει πολύ είναι η κατάχρηση που γίνεται. Μαζί με μένα είναι και ο κύριος Νταλή βέβαια, στον οποίο θα μεταφέρω τις ερωτήσεις σας για το αλκοόλ και τις διαφημίσεις. Πιο συγκεκριμένα αυτός που ασχολείται ε, με αυτή την πτυχή της προστασίας των καταναλωτών θα τα δει. Συνεργαζόμαστε πολύ πάντως και για την Single Market Act με τον κύριο Νταλή. Κυρία Μαριάννα Κογιά, ξέρετε ότι Όλες οι πτυχές της ενιαίας αγοράς με ενδιαφέρουν πολύ και αυτό της κοινωνικής συνεργασίας όλος ιδιαίτερος. Πολύ χάρηκα με την επιτυχία που είχε διάσκεψη που οργάνωσε Κομισιόν με τον κύριο Αντόρ και τον κύριο Ταγιάννη την Παρασκευή. Ο καθηγητής Γιουνούς ήρθε και μίλησε και ο κύριος Μπαρόσο και πολύ. Ήταν ε, Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που ακούσαμε. Υπάρχει και η πρόταση για το νέο μηχανισμό αλληλεγγύης που θα τον έχουμε το 2012, αλλά δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα του 2012 γιατί θα ανακοινωθεί φέτος ακόμα, μέσα στο 2011. Και θα υπάρξουν και άλλες προτάσεις που έχουν να κάνουν με τα θέματα του ε, καταστατικού, των ε, ασφαλίσεων, το θέμα επίσης των πιστοποιητικών για τις αλληλέγγυες επιχειρήσεις ή για τις ηθικές επιχειρήσεις. Πάντως η συνάντηση αυτή η διάσκεψη που είχαμε την ε, Παρασκευή πολύ βοήθησε. Κυρία Κορατσαβίλ, για το ψηφιακό χαρακτήρα. Δεν υπάρχει μία μόνο λύση, ιδιαίτερα για τα προβλήματα στα οποία αναφερθήκατε για το copyright. Εγώ επέβαλα ε, μία πρόταση για τα ορφανά έργα. Θα υποβάλω και πρόταση για τα πνευματικά δικαιώματα ε, μέσα στη βδομάδα ακόμα δημιουργού. Δουλεύουμε σημείο προς σημείο έτσι ώστε να καταλήξουμε σε μια ευρωπαϊκή προσέγγιση. Και ξέρω την δυσκολία για το θέμα στο οποίο αναφερθήκατε. Και το iTunes ήταν το Sportify στο οποίο αναφερθήκατε, όντω κολλάει. Το πρόγραμμα δράσης για τις καταχρηστικές εμπορικές αρχές είναι κάτι στο οποίο θα φτάσουμε πριν το καλοκαίρι. Πριν το καλοκαίρι θα έχουμε ένα εργαστήριο γι' αυτό. Αυτός είναι ο στόχος μας και ελπίζω να τον τηρήσουμε. Ο κύριος Μάγερ, όπως και η Μπάρμπαρα Βάιλερ, αναφέρθηκε στο θέμα της εφαρμογής. Το είπα και πριν. Είναι πολύ σημαντικό στα μέσα που έχει η Γενική Διεύθυνση, έχω εδώ τον αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή για την εσωτερική αγορά, τον γνωρίζουν λίγοι από εσά γιατί ανέλαβε πριν από λίγους μήνες. Η κυρία Βάρβαρα. Μέζα αναφερθήκατε σε αυτό. Είναι θέμα αξιοπιστία για μας. Όχι να κάνουμε καινούρια κείμενα, να ετοιμάζουμε καινούριε ρυθμίσει, αλλά να εφαρμόζονται καλά αυτέ που ήδη έχουμε. Πώ λοιπόν θα παρακολουθήσουμε καλύτερα τη σωστή εφαρμογή σε κάθε στάδιο. Πώς θα το πετύχουμε αυτό σε όλες τις χώρες. Εγώ προσωπικά την έχω ξεκινήσει αυτή τη δουλειά. Έχω συναντηθεί με 700 δημοσίους υπαλλήλου. Πολλοί από αυτού δεν είχαν ποτέ δει Ευρωπαίο Επίτροπο. Σε κάθε δηλαδή πρωτεύουσα των χωρών μας οργάνωσα ένα εργαστήριο. Και έφτιαξα κάτι σαν Facebook με τη γενική μου διεύθυνση, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε επαφή με τους 800 περίπου δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι ασχολούνται είτε με τα επαγγελματικά προσόντα είτε με την οδηγία για τις υπηρεσίες και συχνά λέω ότι συνεργαζόμενοι μαζί τους θα καταφέρουμε τα κείμενά μας να ενσωματωθούν σωστά στην εθνική νομοθεσία και να εφαρμοστούν ικανοποιητικά. Η ενσωμάτωση είναι θέμα των κυβερνήσεων. Η σωστή εφαρμογή όμως είναι θέμα των δημοσίων υπαλλήλων. Γι' αυτό λοιπόν θέλω σε προσωπικό επίπεδο αναχώρα μέλος να παρακολουθούμε τη συνέχεια που δίνεται στις οδηγίες μας. Πρέπει να πείσουμε. Μερικές φορές πρέπει να κάνουμε κάτι ακόμα περισσότερο και να μπούμε στη διαδικασία παραβάσεων. Το κάνουμε και με πολλές μεγάλες χώρες όταν πρόκειται για κακή μεταφορά ε, των κοινοτικών οδηγιών στην εθνική νομοθεσία. Το ότι θέλω σε προσωπικό επίπεδο να παρακολουθώ το ότι γίνεται ένα κράτο μέλο είναι κάτι που ισχύει και για τι δημόσιε συμβάσει. Ο κύριο Μέγερ όντω εντόπισε ένα πραγματικό πρόβλημα. Έχουμε ε, με το ένα χέρι το ξύλο με το οποίο να χτυπάμε τα κράτη-μέλη για να φροντίσουν αυτή, αυτός ο νομοθετικός τροχός που γυρνάει εδώ στην Ευρώπη και ο αντίστοιχος τροχός που γυρνάει για την ομοθεσία στα κράτη-μέλη να μην γυρνάνε παράλληλα αλλά ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον. Κάπου να υπάρχει ένας άξονας που τους συνδέει και ο ένας να γυρνάει μαζί με τον άλλον. Αυτό που μας ενδιαφέρει λοιπόν είναι η ποιότητα των ε, κοινοφιλών υπηρεσιών και η ανακοίνωση για την οποία δεσμεύτηκε ο ίδιος ο κύριος Βαρόσο προσωπικά θα παρουσιαστεί πριν τα τέλη του 2011. Το κείμενο το υποβάλλει ο κύριος Αλμούνια και ε, είναι ειλικρούς και μετά θα προχωρήσουμε για τις Γενικές Υπηρεσίες Κοινής Οφειλίας. Υπάρχει βέβαια και το πακέτο για τις δημόσιες αγοράς κείμενο ε, για το οποίο δεσμεύθηκε ο ίδιος ο κύριος Βαρός εδώ μπροστά σας και δουλεύει πάνω σε αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε και Κέμπερ τώρα, μου υπενθύμησε την ανησυχία που μου έχει ήδη αναφέρει και παλιότερα. Ο λόγος ύπαρξης του κειμένου αυτού και είμαι έτοιμο για ό,τι συζητήσεις ε, θέλετε για να το βελτιώσουμε έχει να κάνει με την έλλειψη νομικής ασφάλειας. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να πάνε να δουλέψουν με συμβάσεις παραχώρησης ενθαρρύνονται έτσι και μπορούν πιο εύκολα να κάνουν αυτή την, αυτό το διασυνοριακό άλμα αν γνωρίζουν ποιο είναι το νομικό πλαίσιο. Τώρα για τις παραχωρήσεις δεν, δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο. Ξέρω την ανησυχία σας και εγώ ο ίδιος ήμουνα εκλεγμένος στο τοπικό επίπεδο για 20 χρόνια. Εγώ δεν θα φύγω από τις Βρυξέλλες και θα πάω στις μικρές, στους μικρούς δήμους να τα βάλω ε, για τις, μαζί τους για τις παραχωρήσεις που κάνουν. Όχι. Αλλά υπάρχει ένα χρονικό όριο. Αναφερθήκατε στο όριο. Είναι αλήθεια ότι για να κατασκευαστεί μια γέφυρα, όπως είπατε, χρειάζεται παραπάνω χρόνος. Αν το κάνουμε με σχέση δημοσίου ιδιωτικού, δεν έχουμε όρια στην ε, παραχώρηση αυτή στη σύμβαση παραχώρηση. Ήμουν υπουργό περιβάλλοντος στη χώρα μου και θεωρούσαμε